Good Καλή σας μέρα. Πολύ χαίρομαι που έχουμε μαζί μας τον Φάβιο Μπανέτα, που είναι υποψήφιος για την ε, θέση μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ο, το μέλο Μπενουά Κερέ θα αποχωρήσει από τα καθήκοντά του 31 Δεκεμβρίου 2019 έχοντα ολοκληρώσει 8 χρονη θητεία. Σύμφωνα με το άρθρο 283.2 λοιπόν, της Συνθήκη για τη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωμοδοτεί επί σύσταση του Συμβουλίου όσον αφορά τον ορισμό των ε, μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρική Τράπεζα. 16 Οκτωβρίου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, συζήτησε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον ορισμό του Φάβιο Πανέτα για 8 χρόνια από 1η Ιανουαρίου του 2020. Μετά την σημερινή, μάλλον πριν από τη σημερινή ακρόαση, ο υποψήφιος έλαβε ένα γραπτό ερωτηματολόγιο με 54 ερωτήσεις. Οι απαντήσεις επισυνάπτονται στο σχέδιο σχετικά με τον ορισμό του μέλους. Μετά την ακρόαση θα έχουμε και ψηφοφορία στις 5 σήμερα το απόγευμα, ώστε η Επιτροπή μας να δώσει πρόταση για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί ε, σύστασης του Συμβουλίου. Η ψηφοφορία θα γίνει στις 16 Δεκεμβρίου. Στην αρχή της ακρόασης θα ακούσουμε μια σύντομη εισαγωγή 10 λεπτών από τον υποψήφιο και μετά θα έχουμε ερωτήσεις και απαντήσεις. Οπότε κύριε Πανέτα, έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σε όλους. Θα αναγνώσω την ε, ομιλία μου, αλλά μπορείτε να βρείτε κάποια από τις παραγράφους ε, στη γραπτή εκδοχή για να γλιτώσουμε κάποιο χρόνο. Κυρία Πρόεδρε, μέλη του Κοινοβουλίου, είναι τιμή μου να εμφανίζομαι μπροστά στην Επιτροπή σας. Είναι ένα βασικό βήμα αυτό στη διαδικασία του διορισμού μου ως, ε, στο Διοικητικό Συμβουλίο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είμαι πεπισμένος ότι η λογοδοσία και η διαφάνεια στους πολίτες και τους εκπροσώπους τους είναι απαραίτητη για την λειτουργία της Κεντρικής Τράπεζας. Θέλω πρώτα απ' όλα να αναφερθώ στα επαγγελματικά μου προσόντα και μετά θέλω να αναφέρω και τις απόψεις μου για το τι χρειάζεται για να φέρουμε εις πέρα στις αρμοδιότητες της Κεντρικής Τράπεζας. Επίσης θα αναφερθώ σε κάποιες από τις μελλοντικές προκλήσεις. Έχω υπάρξει ε, μέλο Κεντρική Τράπεζα σε όλο μου τον επαγγελματικό βίο. Άρχισα να εργάζομαι στην Τράπεζα τη Ιταλία το 1985 και έγινα πλήρε μέλο του Συμβουλίου το 2012. Τώρα είμαι από του ε, ε διευθυντέ και πρόεδρο τη ε, Αρχή Εποπτεία των Ασφαλείων στην Ιταλία. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχω συνεισφέρει στη δημιουργία τη Τραπεζική Ένωση ω μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινού Αποπτικού Μηχανισμού από τη στιγμή τη δημιουργία του. Είμαι επίση μέλο του Γενικού Συμβουλίου του ε, Συμβουλίου για τον Συστημικό Κίνδυνο στην Ευρώπη. Ω ε, μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου στην ΕΚΤ έχω υπάρξει σύμβουλο και αναπληρωματικό μέλο από τι αρχέ τη δεκαετία του 2000. Έτσι, έχω δει τα αρχικά χρόνια ε, τη κοινή νομισματική πολιτική και τι δύσκολε στιγμέ τη ε, νομισματική κρίση και τη χρηματοπιστωτική κρίση. Έχω δει επίση τη σημασία τη διεθνού συνεργασία με συμμετοχή σε πολλά διεθνή φόρα. Πάντοτε γνώριζα ότι οι δράσει μα ε, ω μέλη των κεντρικών τραπεζών δεν πρέπει να λαμβάνουν χώρο σε ένα κενό ε, κενό νοήματο. Πρέπει να έχουμε κάποια σοβαρή επιρροή στην καθημερινότητα των ανθρώπων, την αγοραστική του δύναμη, το εισόδημα, τι συντάξει του, την ασφάλεια στην οποία ζουν ε, και τι αποταμιεύσει του. Πρέπει λοιπόν να δράσουμε σε όλα αυτά τα επίπεδα. Βασισμένο στην εμπειρία μου, θα ήθελα να τονίσω τι βασικέ αρχέ που, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να εμπνέουν τι δράσει τη ΕΚΤΕ τα ερχόμενα χρόνια. Πρέπει να ε, φροντίσουμε τη σταθερότητα των τιμών και τη σχετική μας εντολή, επίσης να βασιστούμε σε δεδομένα, να ε, έχουμε μια διαφανή επικοινωνία και να διατηρήσουμε την οικονομική σταθερότητα. Η διατήρηση τη σταθερότητα των τιμών είναι βασική προτεραιότητα για την ευημερία στην Ευρωζώνη. Αυτό είναι και η ουσία τη εντολή μα. Αυτό επιβεβαιώθηκε από όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια τη κρίση, όταν η Ευρωζώνη αντιμετώπιζε τον άνευ προηγουμένου κίνδυνο μια ε, περίοδου διαρκεία με χαμηλό πληθωρισμό που θα μπορούσε να οδηγήσει και σε ε, αποπληθωρισμό. Οι κίνδυνοι για τη σταθερότητα των τιμών πήγαιναν χέρι-χέρι με τη χαμηλή ανάπτυξη, την, την χαμηλή απασχόληση και το τέλμα στι τιμέ καθώ και τι απειλέ στην ε, χρηματοοικονομική σταθερότητα. Αντιμετωπίσαμε αυτέ τι ε, δυσκολίε όπως τον αποπληθωρισμό, την τάση ε, της ε, επιδείνωσης και της υποβάθμισης με τον πληθωρισμό. Η εμπειρία μας έδειξε ότι όταν αναλαμβάνουμε δράση προτού αποπληθωρισμός οδηγήσει τους οικονομικούς, φορούς να καθυστερι... οικονομικούς φορείς να καθυστερήσουν αγορές και επενδύσεις, είναι σημαντικός τρόπος για την καταπολέμησή του. Έτσι, ε, η αναχέτηση του αποπληθωρισμού βοήθησε την ανάπτυξη και την απασχόληση. Η οικονομία της Ευρωζώνης αντιμετωπίζει ακόμα δυσκολίες λόγω των διεθνών εντάξεων τάσεων και των τάσεων προστατευτισμού. Ε, με την ε, ε, σταθερότητα των τιμών να απειλείται, καθώ και την οικονομική δραστηριότητα να αποδυναμώνεται. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτού του κινδύνου και ταυτόχρονα πρέπει να βρισκόμαστε σε επαγρύπνηση για τι απρόσμενε συνέπειε τη νομισματική πολιτική, ιδίω στην περιοχή τη χρηματοοικονομική σταθερότητα. Ένα υψηλό επίπεδο επιφυλακή είναι απαραίτητο για να δούμε τι συνέπειε που μπορεί να προκύψουν όσο το δυνατόν νωρίτερα. Η Τα εργαλεία μακροπροληπτική πολιτική είναι διαθέσιμα και θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε για να μην υπάρξουν παρενέργειε. Η νομισματική πολιτική δεν μπορεί να ακολουθεί μια προδιαδιαγραμμένη πορεία. Τα μέλη των κεντρικών τραπεζών πρέπει να είναι ρεαλιστέ και να βασίζονται σε δεδομένα για να χρησιμοποιούν διαρκώ ό,τι νέε πληροφορίε προκύπτουν. Η πείρα μου ω ε, οικονομολόγο στην πράξη, καθώ και ο επαγγελματικό μου βίο στην Τράπεζα τη Ιταλία, μου δίδαξαν ότι πρέπει να έχουμε μια ανοιχτόμυαλη αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων. Να παραθέσω και μια δήλωση του πρώην διευθυντή τη Τράπεζα τη Ιταλία και πρώην Προέδρου τη ε, Ιταλική Δημοκρατία Τσάμπη, που είπε ότι το να συγκεντρώνει κανεί γνώση συγκεντρώνοντα αποδεικτικά στοιχεία και να έρχεται αντιμέτωπο με αμφιβολίε, είναι κάτι που επιτρέπει να λαμβάνει κανεί ε, τεκμηριωμένο συγκεκριμένε αποφάσεις. Έτσι, η ανοιχτόμυαλη προσέγγιση για τα εργαλεία μα με, με διαλλακτικότητα σημαίνει ότι ακολουθούμε σωστά την εντολή μα. Τα νέα εργαλεία μπορεί να δημιουργήσουν επιθύμητες παρενέργειε, αλλά η, επιφυλακ... η υπαγρύπνησή μα πρέπει να είναι σε ψηλά επίπεδα. Σε αυτή τη συγκυρία θα πρέπει να εξοπλίσουμε τι πολιτικέ τη ΕΚΤ για να μην υπάρξουν τέτοιε παρενέργειε. Και βεβαίω δεν μπορούμε να ε, παραμείνουμε και να επαναπαυτούμε στι ε, δάφνε μα. Ε, η ξεκάθαρη και διαφανή επικοινωνία είναι, είναι ε, προτεραιότητα για να έχουμε μια αποτελεσματική λειτουργία και να προσανατολίσουμε τι αντιδράσει των αγορών και των πολιτών εκεί που πρέπει. Είναι επίση προπόθεση ώστε οι κεντρικέ τράπεζε να μπορούν να λογοδοτούν στο δημοκρατικά εκλεγμένα σώματα. Αυτό είναι σημαντικό σε στιγμές κρίσης, ιδίως όταν μέτρα αντισυμβατικά πρέπει να εξηγηθούν στο κοινό με σαφήνεια και με σαφή αναφορά στην εντολή για τη σταθεροποίηση των τιμών. Από την αρχή τη κρίση, η Τράπεζα τη Ιταλία ενίσχυσε την επικοινωνία τη και τη λογοδοσία τη προ τη Βουλή. Και από το 2014 το Συμβούλιο έχει εμφανιστεί σε 38 ακροάσεις. Επιπλέον, έχουμε ξεκινήσει ένα πλούσιο πρόγραμμα για να ε, έρθουμε σε επαφή με όλους τους χώρους της κοινωνίας ο ίδιος εγώ έχω συμμετάσχει σε συναντήσεις με πολίτες από διάφορες ιταλικές πόλεις για να συζητήσουμε τις πολιτικές μας και αυτές του ευρωσυστήματος. Αυτό θα βελτιώσει την κατανόηση του κόσμου και την εμπιστοσύνη τους. Η ΕΚΤ έχει βασικές ε, ευθύνες ό,τι αφορά την ε, οικονομική σταθερότητα. Και αυτό γιατί είναι προπόθεση για την σταθερότητα του τιμών, αλλά όχι μόνο. Ω μέλο του Εποπτικού Συμβουλίου ασχολήθηκα με την αρνητική κληρονομιά τη κρίση, για να το πω έτσι. Έξι χρόνια μετά τη δημιουργία του κοινού εποπτικού μηχανισμού, το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα είναι πιο ανθεκτικό, περισσότερο κεφαλαιοποιημένο και καλύτερα εξοπλισμένο για να αντισταθεί σε κλειδονισμούς. Στην Ιταλία ε, τα μη αποδίδοντα δάνεια είναι κάτω από το 4% λιγότερο από την ύψιστη αξία του το 2015. Οι κίνδυνοι τώρα μπορεί να σωρεύονται για μερικούς ε, διαμεσολαβητές εξωτραπεζικούς καθώς και εταιρείε ή τον τομέα των χρηματομεσητικών. Αυτό πρέπει να το παρακολουθούμε στενά με μακροπροληπτικά μέτρα, προκειμένου να ενισχύσουμε την αντοχή τη Ευρωζώνη σε περίπτωση μελλοντικών τριγμών. Πρέπει να υπάρξει πρόοδο στην Τραπεζική ε, Ένωση, ιδίω στον τρίτο πυλώνα, το κοινό σύστημα εξασφάλιση των καταθέσεων, καθώ και την Κεφαλαιοχική Ένωση. Πρέπει τα δύο αυτά προγράμματα να προχωρήσουν για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση και την ευρωστία τη. Ε, για να δούμε τι μελλοντικέ προκλήσει τώρα. Η ψηφιοποίηση αλλάζει τι ζωέ του κόσμου. Η ε, η διείσδυση της τεχνολογίας στα χρηματοοικονομικά πρέπει να γίνει με τρόπο φτηνό, ταχύ και να υπάρξουν ασφαλείς υπηρεσίες για τον ανταγωνισμό και την συμμετοχή όλων στα χρηματοοικονομικά βελτιώνοντας την ευημερία του κόσμου. Αυτό όμως δημιουργεί και δυσκολίες, διότι κάποια, όπως η προστασία των καταναλωτών, είναι εκτός της εντολής της ΕΚΤ. Παρ' όλα αυτά, οι κεντρικέ τράπεζε είναι ζωτική σημασία για να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση στο μελλοντικό ε, τοπίο πληρωμών ε, οι κεντρικέ τράπεζε οι ίδιε πρέπει να υιοθετήσουν νέα τεχνολογικά μέσα. Η Τράπεζα τη Ιταλία έχει αρχίσει να, χρησιμοποιήσει, να χρησιμοποιεί τη μηχανογραφημένη εκμάθηση και τι τεχνολογίε μεγάλων δεδομένων εδώ και χρόνια. Θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά για τι μακροοικονομικέ μα προβλέψει, για να εντοπίζουμε τι ε, παράτυπε συναλλαγέ, καθώ και του δείκτε ε, κινδύνου πραγματικού χρόνου. Θα πρέπει να φροντίσουμε να αντιμετωπίσουμε τι δυσκολίε του μέλλοντο με του μεγάλου άλλου ομίλου, για τι τράπεζε, για την φορολογική συμμόρφωση, για του ε, καταναλωτέ, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την καταπολέμηση τη τρομοκρατία, την νομισματική πολιτική και την χρηματοοικονομική σταθερότητα. Θα πρέπει να υπάρξει ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ δημοσίων αρχών, μεταξύ άλλων και των κεντρικών τραπεζών. Οι εκθέσει για, τα διεθνή, για, τις διεθνή, για τα διεθνή ψηφιακά νομίσματα από την ομάδα εργασία των αναπληρωτών του G7, τον, το οποίο έχω υπάρξει μέλο, ε, προσφέρει σχετικέ ε, μελέτε και αναλύσει. Επίσης οι κλιματικές αλλαγές είναι μια μελλοντική πρόκληση. Θα πρέπει ε, να δούμε και πώ θα επηρεάσουν τη χάραξη πολιτική και την χρηματοοικονομική σταθερότητα. Από αυτή την άποψη, οι κεντρικέ τράπεζε έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν και μπορούν ε, και οφείλουν να αναλάβουν το μερίδιο τη ευθύνη του στην Τράπεζα τη Ιταλία έχουμε κινηθεί προ αυτή την κατεύθυνση. Ω πρόεδρο τη Επιτροπή Επενδύσεων, έχω διευθύνει την ε, ε, επενδυτική μα πολιτική προ την ε, συμπερίληψη αυτών των μερευνών στην δημιουργία του χαρτοφυλακίου επενδύσεών μα, αποκλείοντα εταιρείε που δεν ικανοποιούν τα κριτήρια του Διεθνού Συμφώνου του ΟΗΕ και που έχουν επίση συμπεριλαμβάνοντα αυτέ που έχουν υψηλά περιβαλλοντικά, περιβαλλοντικές επιδόσεις. Θα πρέπει να ενισχύσουμε το δίκτυο για το πρασίνισμα στο χρηματοοικονομικό σύστημα σε διεθνέ και εθνικό επίπεδο με τι σχετικέ τεχνικέ ομάδε. Θα πρέπει επίση η ταξονομία για τι πράσινε δραστηριότητε, να γίνει ένα στόχο που θα επιτρέψει στις σχετικές, ε, στα σχετικά αξιόγραφα και τι κεντρικέ τράπεζε, να διευθύνουν ε, αναλόγω τι δραστηριότητέ του. για περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα. Οι κεντρικέ τράπεζε μπορούν να έχουν καταληπτικό ρόλο στην επενδυτική πολιτική του ιδιωτικού τομέα. Θα πρέπει να ενθαρρύνουν του ε, μεσολαβητέ να συμπεριλάβουν του κλιματικού ε, κινδύνου και τι ε, κοινωνικέ μέρημνε στι πολιτικέ του. Θα πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε και να τονίσουμε τα ωφέλη τη ποικίλη και ε, συμμετοχική διαδικασία λήψη αποφάσεων. Θα πρέπει ε, σε έναν κόσμο παγκοσμιοποιημένο, με τόσο έντονη ε, επικοινωνία, να έχουμε και καλύτερε επιδόσει. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τι διαφορετικέ πτυχέ τη ποικιλομορφία. Την ποικιλομορφία στην σκέψη, στην παιδεία και κυρίω στα φύλλα. Η Τράπεζα της Ιταλίας άρχισε να ασχολείται με την ισότητα των φύλων εδώ και χρόνια, υιοθετώντα ε, ένα πολιτέ στρατηγικό πρόγραμμα και δημιουργώντας και ορίζοντας μάλλον, διορίζοντας έναν μάνατζερ για την ε, ποικιλομορφία, συμπεριλαμβάνοντας πολιτικές και για την ε, επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών. Η ευφυής εργασία και η διαθεσιμότητα μεριμνών ε, δομών παιδική μέρημνα βοήθησε την εξισορρόπηση επαγγελματικού και κοινωνικού βίου, κυρίως για τι γυναίκε. και αυτό είναι σημαντικό. Σε όλα τα πάνελ πρέπει να υπάρχει ισότητα των φύλων και να αποκλείεται η διακριτική μεταχείριση. Τα αποτελέσματα είναι αυτά. 30% των μάνατζερ στην τραπεζά μα είναι τώρα γυναίκε τουλάχιστον ε, πάνω από το μισό σε σχέση με τα περασμένα χρόνια. Έχουμε ξεπεράσει το στόχο του 35% μέχρι το 2022 και θα συνεχίσουμε να ε, κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Για την αρχή εποπτείας των ασφαλιών στην Ιταλία, όπου είμαι πρόεδρος, οι γυναίκες σε θέσεις μάνατζερ είναι 50%. Ε, η ισότητα των φύλων ω προ την εκπροσώπησή μα ε, στα διάφορα επίπεδα, καθώ και τι φωνέ που ακουγόνται στη τραπέζια των διαπραγματεύσεων, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να επιδιώκει η ΕΚΤ. Να ολοκληρώσω λέγοντα ότι έχω δει πόσο αφοσιωμένη είναι η Επιτροπή σα ε, στην εξέταση των θεμάτων που ανέφερα. Η συζήτηση και η εξέταση τέτοιων θεμάτων από το Ευρωκοινοβούλιο είναι πραγματικά ε, ένα σημαντικό στοιχείο για την αποτελεσματική λειτουργία τη ΕΚΤ. Πιστεύω ότι οι οικονομικέ ε, και χρηματοπιστωτικέ μου γνώσει, καθώ και η εμπειρία μου, μπορούν να συνεισφέρουν στην ολοκλήρωση τη εντολή τη ΕΚΤ και στην αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων. Ως εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών, εσείς ε, είστε υπεύθυνοι για την επιλογή μου και θα είναι τιμή μου να με υποστηρίξετε εάν διοριστώ στο Διοικητικό Συμβούλιο του ε, ΕΚΤ. Έτσι θα μπορέσω και εγώ να συμβάλλω στην ε, οικοδόμηση μιας ισχυρότερης και συμμετοχικότερης καθώς και πιο ισότιμης Ευρώπης. Σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Αρχίζουμε τώρα με ερωτήσεις και απαντήσεις. Πέντε λεπτά για τον καθένα. Και αρχίζουμε με τον κύριο Μάρκες από το ΕΛΚ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πανέτα, αν μου επιτρέπετε θα μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα. Είπατε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν με ευέλικτο τρόπο τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας και μιλήσατε και για ασυνήθιστα αντισυμβατικά μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέχρι τις 31 ε, Δωδεκάτου που δεν είσαστε ακόμη εκεί ε, θα έχει εξαντλήσει τα μέσα για να αντιδράσει σε ε, αρνητικές οικονομικές τάσεις. Η πρόεδρος, η κυρία Λαγκάρτ είπε ότι δεν θα επιτρέπεται να περιορίσουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε, να απαγορέψουμε διάφορους τρόπους σκέψης. Εσείς ε, τι εννοείτε, αγορά ε, μετοχών, ε, κατάργηση των μετρητών ή έχετε άλλες ιδέες στο νου σας. Καταρχάς, σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας που θίγει ένα πολύ σημαντικό θέμα. Εγώ αναφερόμουν σε οποιοδήποτε μέσο, συνηθισμένο ή ασυνήθιστο. Ε, όπως ξέρετε, η ασυνηθιστο οπως ξερετε η θεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχει αλλάξει ε, για να πετύχει τον στόχο της, του πληθωρισμού. Πέρασε λοιπόν από συνηθισμένα μέτρα σε μη συνηθισμένα μέτρα, όπως είναι το πρόγραμμα αγοράς ε, ε, περιουσιακών στοιχείων ε, ή τα αρνητικά επιτόκια. Αυτό ήταν απαραίτητο διότι ε, έπρεπε να αντισταθμίσουμε τον κίνδυνο ε, ε, ενός σπιράλ πληθωρισμού ή τώρα που έχουμε, από ό,τι φαίνεται, μια μακρά περίοδο σταθερότητας. Δεν σκέφτομαι τα χρήματα ελικόπτερο, όπως λέμε, τα, τις ξαφνικές χρηματοδοτήσεις. Σκέφτομαι όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να διατηρήσει τη σταθερότητα των τιμών. Ας σκεφτούμε πώς είχε η κατάσταση πριν 10 χρόνια. Ποιος μπορούσε τότε να φανταστεί ότι σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αγόραζε ομόλογα με αρνητικά επιτόκια ή σε άλλες δικαιοδοσίες ότι ε, η Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών θα εφήρμοζε τα μέτρα που εφηρμάζει ή ότι η Ιαπωνία θα ξεκινούσε ποσοτική χαλάρωση ε, αγοράζοντας και μετοχές μη χρηματοοικονομικών εταιριών. Δεν είναι κάτι δεν έχουμε κατά νου τέτοια μέτρα, αλλά φαίνεται έτσι η ανάγκη για λήψη μέτρων αναλογικών και απαραίτητων για να διατηρήσουμε τη σταθερότητα των τιμών. Επιτρέψτε μου μία συμπληρωματική ερώτηση. Ο Μάριο Ντράγη είπε στην τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Τράπεζας ότι δεν ήταν ανάγκη να γίνει ψηφοφορία διότι ήταν σαφής η πλειοψηφία. Εκ των υστέρων φάνηκε ότι δεν ήταν καθόλου τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα και ότι υπήρχαν ε, σημαντικές ε, αντιρρήσεις από μια σειρά κρατών μελών. Εσύ πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να βελτιωθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων ε, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και πώς βλέπετε το δικό σας ρόλο στη διαδικασία αυτή. Δεν συμμετείχα στην ε, συνεδρίαση αυτή, ε, οπότε θα σας απαντήσω με βάση τις δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες. Οι πληροφορίες που έλαβα Ε, και σχετικά με τα όσα είπε η πρόεδρος του, ε, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας χθες, ε, φαίνεται ότι υπάρχει ανάγκη για ομοφωνία όσον αφορά την ανάγκη ε, για μέτρα μεγέθυνσης επεκτατικής πολιτικής. Και Συμμετείχα σε προηγούμενες συνεδριάσεις ε, του Διοικητικού Συμβουλίου, ε, οι οποίες πάντα ξεκινούν με μια πολύ αναλυτική παρουσίαση των οικονομικών εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο, ε, στην Ευρωζώνη, την κατάσταση των χρηματοοικονομικών αγορών. Και η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι πολύ τεχνική πολλές πληροφορίες δίδονται και γενικά πιστεύω ότι τα μέλη του Συμβουλίου θεωρούν κατάλληλη την όλη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Σε ένα Συμβούλιο με 25 μέλη δεν θα πρέπει να εκπλήσει κανέναν αν ιδιαίτερα σε ε, ιδιαίτερες καταστάσεις όπως η παρούσα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, υιοθέτησε ε, μια δέσμη μέτρων που δεν ε, ανήκουν στη συνηθισμένη εργαλειοθήκη των κεντρικών τραπεζών και σε μια τέτοια περίπτωση να υπάρχουν και διστάμενες απόψεις. Αλλά μέχρι τώρα η διαδικασία λήψη αποφάσεων έχει φανεί αποτελεσματική και το Διοικητικό Συμβούλιο πάντα μπορούσε να λάβει αποφάσεις και να επέμβει εν οπότε αυτό ήταν απαραίτητο. Σας ευχαριστώ. κύριος Φερνάντες από τους Σοσιαλδημοκράτες. Καλή σας ε, μέρα. Θα μιλήσω ισπανικά. Καλώς ήρθατε κύριε Πανέτα. Δύο ερωτήσεις έχω παρακαλώ. Όπως γνωρίζετε γίνεται ακαδημαϊκή συζήτηση σχετικά με την εξέλιξη των φυσικών επιτοκίων στο βαθμό που υπάρχει μια μόνιμη μείωση των ε, επιτοκίων αυτών. Οπότε θα ήθελα να ξέρω στα πλαίσια της αναθεώρησης του πλαισίου της νομισματικής πολιτικής που ζήτησε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την ακρόαση που είχε με την κυρία Λαγκάρτ και που χτες μας ανακοίνωσε επίσημα εδώ η κυρία Λαγκάρτ, θα ήθελα να γνωρίζω σε τι βαθμό η αναθεώρηση αυτή μπορούμε να πούμε ότι θα ασχοληθεί με τα φυσικά αυτά επιτόκια έτσι ώστε να υπάρξει αλλαγή και όσον αφορά τον στόχο του πληθωρισμού. Δεύτερον, όλοι ανησυχούμε, όπως είπατε κι εσείς, για τις παρενέργειες της ε, τρέχουσας νομισματικής πολιτικής. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου πιστεύετε ότι θα μπορούσε να είχε καλύτερο ρόλο στον σχεδιασμό των μακροπροληπτικών ε, πολιτικών έτσι ώστε να περιοριστούν αυτές οι παρενέργειες. Ευχαριστώ. Απάντηση. Σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, όπως ανακοίνωσε η Πρόεδρος, το Συμβούλιο Δικητών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα συζητήσει την στρατηγική νομισματικής πολιτικής. Έτσι λοιπόν η προσέγγιση θα είναι μια ευρεία προσέγγιση και οι συζητήσεις θα γίνουν συνολικά. Υπάρχουν πολλά και διαφορετικά στοιχεία της νομισματικής πολιτικής που θα ληφθούν υπόψη. Έχετε δίκιο πάντως ε, στον εκαθημαϊκό κόσμο. Ένα από τα πράγματα με τα οποία συμφωνούν οι εμπειρογνώμονες, οι οικονομολόγοι, είναι ότι τα φυσικά επιτόκια μειώνονται εξαιτία των παγκοσμίων τάσεων της περιορισμένης ε, μεγένθησης, των ε, αποταμιεύσεων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα άρθρα τα οποία προτείνουν για να απαντήσουμε σε αυτήν την μείωση αρκεί να αλλάξουμε τον στόχο μας για τον πληθωρισμό. Κάποιοι βέβαια στα άρθρα τους λένε ότι πρέπει να αυξηθεί, αυτός ο στόχος άλλοι λένε να μειωθεί. Είναι πράγματα τα οποία θα συζητήσει σίγουρα το Συμβούλιο Δίκητων. Θα κάνει την κατάλληλη ανάλυση και με τη βοήθεια και ακαδημαϊκών απ' έξω, ε, τα μέλη της κοινωνίας, Εβραίος κλπ. Σίγουρα και άλλα στοιχεία θα συζητηθούν εν ώψη της αναθεώρησης αυτής της στρατηγικής μας για την νομισματική πολιτική. Έρχομαι στη δεύτερη ερώτησή σας τώρα. Ναι, υπάρχουν παρενέργειες. Όσον αφορά τα μέτρα αυτά πολιτικής και νομίζω ότι οι παρενέργειες αυτές έχουν εντοπιστεί από, τη, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου που εξέδωσε και προειδοποίησεις πολλές φορές, σε πολλές περιπτώσεις, όταν υπερθερμάθηκε ας πούμε η αγορά στέγασης. Και σε πολλές χώρες εντοπίστηκε αυτό το πρόβλημα και αναλύθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου. Τώρα πιστεύω ότι στην Ευρωζώνη υπάρχουν 13 χώρε οι οποίες έχουν υιοθετήσει μακροπροληπτικά μέτρα για να αντιμετωπίσουν ακριβώς την αύξηση των τιμών τη στέγαση. και οι προειδοποίησει αυτές και αυτά τα μέτρα μάλλον, τα μακροπροληπτικά, ε, προχώρησαν μετά από σύσταση ακριβώς δικιά μας. Οπότε, είναι ο κατάλληλος χώρος για να εξετάζονται οι επιδράσεις της νομισματικής πολιτικής και μακροπροληπτικά και γενικότερα. Είναι μια πάρα πολύ πολύτιμη συνεισφορά στη νομισματική πολιτική της ε, Ευρωζώνης. Ευχαριστούμε. Η Μόνικα Σενλέπο τώρα, από το Ρινιού. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πανέτα. Την προηγούμενη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία υπερψήφισε το ψήφισμα ε, για το κλίμα. Σημαντικό μήνυμα προς τους πολίτες μας αλλά και προς όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι θα πρέπει να αναλάβουμε επιγόντως δράση. Η επανεξέταση τη νομισματική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι τώρα το θέμα μα και η κυρία Λαγκάρντε στην επιτροπή μα χθε ε, είπε ότι, θα πρέπει, ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης ε, κριτήρια κλιματικά. Και εσείς ε, στην εισήγησή σας και στην εισήγησή της είχε αναφερθεί σε αυτό. Εσείς πιστεύετε ότι η αλλαγή του κλίματος ή η ψηφιοποίηση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ε, κατά τη δημιουργία ενός πιθανού ψηφιακού νομίσματος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, διότι δεν φαίνεται όλα τα μέλη του Συμβουλίου να συμφωνούν με κάτι τέτοιο. Ε, επικεντρώνονται αποκλειστικά σε θέματα ε, χρηματικά, νομισματικά. εσείς πώς το βλέπετε. Δύο ερωτήσεις κατάλαβα ότι μου θέτετε. Η πρώτη έχει να κάνει με τη σχέση ανάμεσα στις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και την αλλαγή του κλίματος. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει τρία καθήκοντα. Ε, το βασικό είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, κατόπιν ε, είναι η μακροπροληπτική ε, εποπτεία και τρίτον η χρηματοοικονομική σταθερότητα. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην ανάλυση των κινδύνων του κλίματος ε, και με τις τρεις αυτές ιδιότητες ε, και στο πλαίσιο των τριών αυτών καθηκόντων της ε, τράπεζας. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας ήδη έχει ξεκινήσει συζητήσεις με τράπεζες για να τις καλέσει να λάβουν υπόψη και τους κινδύνους από την αλλαγή του κλίματος στις εργασίες τους. Εάν δεν λάβουν υπόψη αυτή την πτυχή μπορεί να υποτιμούν τους ε, κινδύνους που φέρουν. Και θα ήταν καλύτερα μέσω πρόθεσμα να λάβουν υπόψη και τον κίνδυνο από την αλλαγή του κλίματος. Η χρηματοοικονομική σταθερότητα επηρεάζεται και από την ε, ε, αλλαγή του κλίματος. Σκεφτείτε για παράδειγμα τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών σε οικονομικούς φορείς όπως είναι οι ασφαλιστικές εταιρείες κάτι τέτοιο μπορεί τελικά να επηρεάσει και την χρηματοοικονομική σταθερότητα. Και τέλος, στον ε, ρόλο της ε, τράπεζας ε, για την χρηματοοικονομική σταθερότητα θα πρέπει να λάβει υπόψη και, την, και τον κίνδυνο από την αλλαγή του κλίματος. Αλλά πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το θέμα αυτό και στις καθημερινές εργασίες Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, διότι σκεφτείτε το, τις οικονομικές επιπτώσεις ε, ενός πολύ κρύου χειμώνα, για παράδειγμα. Διότι ο χειμώνας εμποδίζει, για παράδειγμα, τις εργασίες στον τομέα των οικοδομών. Μεσοπρόθεσμα, σκεφτείτε τη μετάβαση την ενεργειακή μετάβαση, τον ε, ε, τομέων ε, υψηλής, ε, υψηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Σκεφτείτε τις επιπτώσεις και αυτής της μετάβασης στην οικονομία. Η βασική συνεισφορά λοιπόν της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο περιβαλλοντικό αυτό θέμα είναι να διευκολύνει την τιμολόγηση της αλλαγής του κλίματος όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά ο χρηματοοικονομικός τομέας στο σύνολό του θα χρηματοδοτήσει μέτρα που σχετίζονται με θέματα περιβαλλοντικά. Υπάρχει η δυνατότητα της Κεντρικής Τράπεζας επίσης να επενδύει τους δικούς της πόρους ε, στην αγορά κινητών αξιών ε, φιλικών προς το περιβάλλον. Πρόκειται για τα λεγόμενα πράσινα ομόλογα. Αλλά θα πρέπει να λάβει κανείς υπόψη και την ανάγκη ουδετερότητας ως προς ε, την αγορά της ε, Κεντρικής Τράπεζας. Αυτές οι επενδύσεις ε, μάλλον θα συνεχίσουν να αυξάνονται όσο αυξάνεται και η αγορά συγκεκριμένα νούμερα. Σύμφωνα με διεθνή οργανισμό υπάρχουν 7 δισεκατομμύρια πρασίνων ομολόγων. Εξ αυτών ε, μόνο τα 250 εκατομμύρια βρίσκονται στην Ευρωζώνη. Ας σκεφτούμε ότι το μισό αυτών βρίσκεται στα χέρια επενδυτών. Ε, αυτό σημαίνει ότι μόλις πάνω από 100 δισεκατομμύρια ε, πράσινων ε, επενδύσεων είναι διαθέσιμο. Εάν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μόλις το 5% διέθετε σε πράσινα ομόλογα θα καταβρόχθιζε το σύνολο της αγοράς στον τομέα αυτών. Πρέπει λοιπόν να είμαστε προοδευτικοί. Δεν θέλουμε να αφαιρέσουμε ρευστότητα από την αγορά, δεν θέλουμε να καταστήσουμε αδύνατο σε ιδιωτικού ε, επενδυτέ να ε, επενδύουν ε, σε πράσινα ομόλογα. Ευχαριστώ πολύ, Γιακοπιούνας, από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ πολύ. Είναι σημαντικές όλες αυτές οι προκλήσεις που αναφέρετε. Ας προσπαθήσουμε όμως να πάμε λίγο περισσότερο σε βάθος. Δεν θα συμφωνούσατε ότι ο τραπεζικός τομέας είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα παρά την όποια επέκταση. Το θέμα της δημιουργίας χρήματος, της νομισματικής πολιτικής, σε ένα μεγάλο βαθμό τουλάχιστον, όπως επίσης οι αναντιστοιχίες των ισολογισμών του τραπεζικού συστήματος, γιατί οι τράπεζες πρέπει να αναχρηματοδοτούνται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα όταν φεύγει το χρήμα. Και σε μερικές χώρες είχαμε πρόβλημα το οποίο είναι πολλαπλάσιο του ΑΕΠ μάλιστα. Οπότε το τραπεζικό και το οικονομικό σύστημα γενικό συνδέεται βέβαια και με τις προηγούμενες απορριθμίσεις και τα λεγόμενα, λεγόμενα καινοτόμα προϊόντα. Δεν νομίζετε ότι αυτά είναι τα κύρια προβλήματα που οδήγησαν στην κρίση και μάλιστα όχι μόνο σε αυτή την κρίση αλλά και σε προηγούμενες. Οπότε ποια είναι η γνώμη σας για αυτές τις δηλώσεις. Συμφωνείτε σε ένα βαθμό ε, πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στο τραπεζικό σύστημα και τους διάφορους μηχανισμούς ώστε να αντιμετωπιστούν ακριβώς αυτές οι προκλήσεις που δεν ήρθαν για να φύγουν γρήγορα δυστυχώς. Οπότε, ό,τι προγράμματα υπάρχουν για τις ε, τράπεζες σίγουρα θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Απάντηση. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Είναι αλήθεια ότι το μοντέλο fractional reserve είναι ασταθές. Και ξεκίνησε πριν από την οικονομική κρίση. Μετά τη Λίμαν, οι ρυθμιστικές αρχές αντέδρασαν. Και κάποιοι νέοι νόμοι αποφασίστηκαν και άλλαξε βέβαια και η εποπτική προσέγγιση. Θα λέγαμε μάλιστα σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπήρξαν μέτρα τα οποία λήφθησαν για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα ζητήματα που αναφέρατε, η αναντιστοιχία με θέματα ληκτικότητας πώς να προστατεύεται η τράπεζα από πρόβλημα έλλειψης ε, ρευστότητας αν ε, πρέπει να δώσουν το έχουν θέμα με το παθητικό τους. Τώρα λοιπόν είναι πιο συντηρητικά τα μέτρα, είμαστε πιο προσεκτικοί και θα πρέπει να υπάρχει και, ένα, ε, και μια μόχλευση σε σχέση με το σύνολο του ενεργητικού των τραπεζών το απόθεμα δηλαδή των τραπεζών, η κεφαλοποίησή του να είναι επαρκή. Αυτό είναι κάτι που επίση έχει αλλάξει. Αντιμετωπίστηκαν λοιπόν αυτά τα ζητήματα μετά την κρίση. Τώρα στην Ευρωζώνη η αντίδραση ήταν έντονη μετά την κρίση. Ξεκινήσαμε με τον ενίο εποπτικό μηχανισμό και ήδη έχουμε τον πρώτο πυλώνα που λειτουργεί με αποτελέσματα εποφελή ε, και που τα βλέπουμε ήδη όσον αφορά την εποπτεία. Είπα εισαγωγικά για το λόγο των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς τα συνολικά δάνεια και έχει μειωθεί ο λόγος αυτός. Υπάρχει απομόχλευση επίσης στις τράπεζες. Ε, το σύνολο του ενεργητικού σε σχέση με το ΑΕΠ έχει μειωθεί. Και επίσης έχουν εισαχθεί και διάφορες ρήτρε για να ελέγχεται ο κίνδυνος ε, του τραπεζικού συστήματος. Υπάρχει βέβαια και ο νέος υποπτικός, ε, μάλλον το, υπάρχει το ενιαίο Συμβούλιο Εξυγένσης τώρα που επίσης αρχίζει να λειτουργεί και έχει ήδη παρέμβει σε μερικές περιπτώσεις κρίσης τραπεζών. Και έχει λειτουργήσει και αρκετά καλά αυτός ο μηχανισμός. Το ζήτημα είναι ο τρίτος πυλώνας τώρα που θα έπρεπε να ε, εισάγει την, ε, τις εγγύσεις καταθέσεων. Οι συζητήσεις από αυτού συνεχίζονται. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μετά από το γερμανικό non-paper για την ε, Τραπεζική Ένωση. Σίγουρα θα υπάρξουν και άλλες ρήτρες, το backstop, για το ενίο ταμείο εξυγίανσης, το ΤΙΛΑΚ για τις ε, συνολικά συστημικές τράπεζες. Υπάρχουν διάφορες ρήτρε, δηλαδή εξασφάλισης που εισάγονται, που δεν θα έλεγα βέβαια ότι αποκλείουν, αλλά τουλάχιστον ελέγχουν το τραπεζικό σύστημα ώστε να μην κινδυνεύει η οικονομία από αυτό. Αντώνιο Ρινάλντι τώρα, ID. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πανέτα, με τέτοιο επαγγελματικό προφίλ στις κορυφές της πιο γνωστής τραπεζικής αρχής της Ιταλίας, την ε, Τράπεζα της Ιταλίας. Δεν θεωρείτε ότι είναι ένα σοβαρό προσόν για το διορισμό σα στο Διοικητικό Συμβούλιο τη ΕΚΤ. Παρ' όλα αυτά, έχω κάποιε ερωτήσει. Νομίζετε ότι οι αρμοδιότητε του Μηχανισμού Σταθερότητα θα πρέπει να είναι μέρο τη εντολή τη ΕΚΤ, όπω όλε τι κεντρικέ τράπεζε του κόσμου, και ότι θα πρέπει η πρόληψη του κινδύνου αφαιρεγγιότητας αναχώρα να είναι μέρος των λειτουργιών ε, ε, του, του μηχανισμού αυτού και κατ' επέκταση της Κεντρικής Τράπεζας θα πρέπει να ε, δούμε στο άρθρο 3, ε, εδάφιο 1 του ιδρυτικού κανονισμού της ΕΣΜΑ, τι γίνεται με τη μακροοικονομική κατάσταση των κρατών μελών και κατά πόσον η βιωσιμότητα του χρέους ασχέτως της ενεργοποίησης του μηχανισμού μετά από αίτημα του κράτους ε, ε, περιλαμβάνει την δυνατότητα εισαγωγής βαθμολόγησης ε, επιδόσεων. Αυτό μπορεί να είναι καταστροφικό σε περίπτωση Αυτό θα πρέπει να ε, ληφθεί υπόψη και για να δούμε ποιος πρέπει να καθορίζει αυτές τις επιδόσεις, αλλά χωρίς να πλήξουμε καταστροφικά τις αγορές. Και μετά, σύμφωνα με τη γραμμή του Προέδρου Ντράγκη, για την έκτακτη τόνωση στο, το, της με την ποσοτική χαλάρωση, όπως και γίνεται στο παρελθόν, έχω την εξή ερώτηση. Η ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να λάβουν λιγότερο διακριτικές διευθετήσεις για τις εμπορικές τράπεζες σε αντιδιαστολή με αυτές που έχουν χρηματοοικονομικές δραστηριότητες και κυρίως διευκολύνσεις για παράγωγα και derivatives τα οποία είναι το επίπεδο 3. Ε, θα δούμε λοιπόν και σας εύχομαι καλή δουλειά. Thank you very much for your... Ε, Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Να απαντήσω τελικά. Μπορώ και στα αγγλικά βέβαια. Πρώτα απ' όλα για τον ειδικό κανονισμό του ESM, του Μηχανισμού Σταθερότητας. Θεωρώ ότι ο κανονισμός αυτός ορίζει την νομική βάση για τη λειτουργία του ESM και την δίκησή του ως οργάνου. Δεν βλέπω να υπάρχουν μείζονο σημασία αλλαγέ ε, με την αλλαγή του κανονισμού. Ε, χρειάζεται εδώ λοιπόν μια πολιτική ασφάλειας για να το πω έτσι. Μια ασφάλεια που ε, όλοι τη θέλουμε και την αγοράζουμε ελπίζοντας ότι δεν τη χρειαστούμε ποτέ. Όπω και σε ένα ατύχημα. Δεν ελπίζουμε να έχουμε ατύχημα για να χρειαστούμε την ασφάλεια, αλλά έτσι ισχύει και για τον ΕΣΜ, τον ESM. Εδώ λοιπόν σκοπό έχει να ενισχύσει τη δυνατότητα αντιμετώπιση κρίσεων της Ευρωζώνης και αυτό είναι και ο στόχος των προτάσεων που βρίσκονται επιτάπητο. Νομίζω ότι αυτή είναι μια καλή στιγμή για να προβλέψουμε αυτό ακριβώς το πλαίσιο. Δεν υπάρχει χώρα η οποία να αντιμετωπίζει χρηματοοικονομικούς τριγμούς Δεν υπάρχει κάποιος που να αντιμετωπίζει πρόβλημα χρέους ε, ή πρόσβαση στι αγορές τι Κανείς δεν έχει πρόβλημα δημόσιου χρέους και δεν υπάρχει χώρα που να μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή που να μοιάζει να είναι σε φάση να, να ανατρέξει στον ESM. Ωστόσο, ε, καλή είναι η στιγμή για να αγοράσει κανείς και την ασφαλειά του τώρα. Εδώ τα μη συμβατικά μέτρα, όπως έλεγα προηγουμένως, μπορεί να χρειαστούν για την σταθεροποίηση των τιμών. Ως τώρα η αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ότι οι προβλέψεις Οι προβλέψεις δείχνουν ότι το 1,5 το 2021 δεν είναι ικανοποιητικό επίπεδο. ώστε να έχουμε μακροπρόθεσμα σταθεροποίηση των τιμών. Το Διοικητικό Συμβούλιο όμω ακριβώς γι' αυτό έλαβε αυτά τα μέτρα το Σεπτέμβριο, γιατί είναι απαραίτητο και ευταίο και να διατηρηθεί αυτή, και αν διατηρηθεί αυτή η συζήτηση, θα λαμβάνουμε αποφασιστική δράση, προκειμένου να δούμε με τι εργαλεία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Για τις τράπεζες είμαι υπέρ του να παρακολουθούμε διαρκώς όλους τους κινδύνους, τις συναλλαγές, τις αγορές, τα e την, ε, την, το ξέπλυμα χανδρόμικου χρήματος, όλα αυτά θα πρέπει να τα έχει υπόψη το μηχανισμός παρακολούθησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Ευχαριστώ. πολύ, Ραφαέλα Φίτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οπωσδήποτε για τους γνώστες του βιογραφικού και της πείρας του κυρίου Πανέτα καταλαβαίνει ότι είστε εγγύηση για τα θέματα που θα μας απασχολήσουν. Εγώ θέλω να κάνω δύο γρήγορες ερωτήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με κάτι που προέκυψε και χθε. Όπως μας είπε η πρόεδρος της ΕΚΤ, στη στρατηγική της αξιολόγηση, τι σκοπεύει να κάνει στο μέλλον. Και εσείς κυρία Πανέτα λέτε ότι η Επιτροπή Στρατηγικής Πολιτικής είναι σημαντική για την μελλοντική σας ε, δράση. Τώρα, ω προς το διορισμό, η στρατηγική μεταρρύθμιση της ΕΚΤ είναι κάτι που έχετε σκεφτεί στι του. Τι μπορείτε να μα πείτε για το τι κατεύθυνση θα πάρει αυτή η μεταρρύθμιση, αυτή η αναθεώρηση. Και κατά δεύτερον, για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Στον ε, τραπεζικό τομέα στην Ευρώπη έχουμε το πρόβλημα της χαμηλή κερδοφορία. Τι θεραπείες, τι μέσα θεραπείε μπορούμε να βρούμε ε, ε, συμπληρωματικά σε σχέση με την αγωγή που έχει δοθεί ήδη μέσα από την εντολή σας για, την, για το περιορισμό του κινδύνου στον τραπεζικό τομέα. Ευχαριστούμε για τις ερωτήσεις σας. Για την πρώτη, για την αναθεώρηση της ε, πολιτικής στρατηγικής στα νομισματικά, σαφώς η αναθεώρηση θα πρέπει να λάβει υπόψη όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν αλλάξει τα τελευταία 15 χρόνια, 16 χρόνια από όταν είχε γίνει η προηγούμενη αναθεώρηση. Έκτοτε άλλαξε εντελώς και η δομή του χρηματο οικονομικού συστήματος. Τα τραπεζικά και εξωτραπεζικά έχουν αλλάξει, οι τράπεζες έχουν αλλάξει τον τρόπο της λειτουργίας τους, οι διαμεσολαβητές ε, που λειτουργούν εξωτραπεζικά έχουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο και είμαστε και σε μια φάση χαμηλής ανάπτυξης με μείωση των πραγματικών ε, επιτοκίων. Οπότε αυτό προφανώς επηρεάζει σε μερικές περιπτώσεις στην Ιαπωνία. Μα αυτά είναι καθιερωμένα πλέον. Γι' αυτό πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί η νομισματική πολιτική. Γιατί θα ήταν περίεργο με βάση τις σημερινές εξελίξεις να μην γίνει. Πρέπει να δούμε ποιο είναι ο καλύτερο δυνατό τρόπο να επιδιώξουμε του στόχου σταθεροποίηση των τιμών. Να δούμε πώ θα διατηρήσουμε τη σταθερότητα των τιμών. Τώρα για την ερώτησή σα για τι τράπεζε. Οι απαντήσει στο ερωτηματολόγιο το λένε. Τόνισα ότι το βασικό πρόβλημα του τραπεζικού τομέα στην Ευρώπη είναι η χαμηλή κερδοφορία. Οι κίνδυνοι που έπληξαν το τραπεζικό τομέα μετά την ε, χρηματοπιστωτική κρίση και όλες τις προσπάθειες που έγιναν δεν λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Τα βασικά συστημικά ζητήματα αντιμετωπίστηκαν από τον νέο μηχανισμό εποπτείας. Και οι συστημικοί κινδύνοι μειώθηκαν στην Ευρωζώνη κατά 50%. Στις χώρες ε, ε, ψηλού κινδύνου η μείωση των εξυπηρετούμενων δανείων ήταν ακόμα πιο μεγάλη. Όμως, υπάρχουν ζητήματα στην αγορά που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Τώρα βλέπουμε όλο ένα και περισσότερε υποθέσει ξεπλήματο βαμικού χρήματο σε ευρωπαϊκέ τράπεζε. Καταλαβαίνουμε ότι ο κίνδυνο του ξεπλήματο χρήματο είναι ένα ύπουλο στοιχείο που μπορεί να φέρει σε δύσκολη θέση την τράπεζα όπω παλιότερα. Τώρα πρέπει να τον ενώσουμε την κερδοφορία των ε, τραπεζών. Το βασικό πρόβλημα που επηρεάζει την κερδοφορία των τραπεζών είναι η δυνατότητα ε, τήρησης περιουσιακών στοιχείων. Αυτό επηρεάζει πιο πολύ. Και υπάρχουν πολλοί τρόποι να το δούμε αυτό. Πρώτα απ' όλα, η εξυγίανση και διασωνηριακά όταν κάνει κανείς μια τέτοια διασυνοριακή εξυγίανση ε, μπορεί να λύσει πολλά ζητήματα χωρίς ε, επιπλέον ε, δυνατότητες στην αγορά και χωρίς να δημιουργήσει προβλήματα εκεί. Αλλά οι τράπεζες πρέπει να αντιμετωπίσουν και τις τεχνολογικές προκλήσεις. Αντιμετωπίζουν τα θέματα ανταγωνισμού, έχουν ανταγωνιστές στην προσφορά συγκεκριμένων υπηρεσιών, τις πληρωμές και τις λόγω χάρη άλλου είδους συναλλαγές ε, από τις λεγόμενες εταιρείες FinTech, αυτές που προσφέρουν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες με πολύ χαμηλότερο κόστος, εξωτραπεζικά. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε το θέμα της υπερδυνατότητας των τραπεζών και να σκεφτούμε πολύ σοβαρά πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τράπεζες που εκτός αγοράς δεν έχουν να κάνουν κάτι άλλο και πώς μπορούμε να τις υποστηρίξουμε πρώτες, δηλαδή να μην έχουν εξωτερικές απώλειες, ε, και να προηγηθούν ε, των ε, συναδέλφων τους χωρίς να χρησιμοποιηθεί το bail-in και bail-out. Αυτό όμως ξέρετε ότι ισχύει για μια χούφτα τραπεζών στην Ευρωζώνη 15-16 Αυτέ έχουν σχέση πιο πολύ και με τα κρατικά συμφέροντα. Όμω για όλε τι υπόλοιπε, 4.000 τράπεζε στην Ευρωζώνη, ξέρετε ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Πέρα από την εξυγίανση, είναι άλλα τα θέματα. Θέματα ρευστότητα και θέματα που θα πρέπει να τα δούμε στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Ρουσμάου τώρα από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω πορτογαλικά Ήθελα να μου πείτε στην αναθεώρηση της στρατηγικής πολιτικής που σκέφτεστε για την νομισματική πολιτική θα δείτε και το θέμα του συνδυασμού της νομισματικής πολιτικής με άλλες οικονομικές πολιτικές. Πιο συγκεκριμένα αυτή του προπολογισμού, τη δημοσιονομική. Και από αυτήν την άποψη πραγματικά μου φαίνεται πολύ ε, ενοχλητικό πώς σκεφτόμαστε όλο ένα και πιο δημιουργικά μέτρα για την νομισματική πολιτική χωρίς να τα συνδυάζουμε και μάλιστα εξισορροπημένα με ε, μέτρα ε, για τον προπολογισμό σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέτρα δημοσιονομικά τα οποία θα μπορούσαν να κατανείμουν καλύτερα τις εκτατικές προσπάθειες. Η απάντηση που παίρνω πάντα όταν θέτω αυτό το ερώτημα σε κάποιον από την Κεντρική Τράπεζα είναι ότι ότι ιδίω στην ΕΚΤ τα θέματα αυτά, η πολιτική του προπολογισμού είναι εκτό τη εντολή τη ΕΚΤ. Αυτό όμω προκαλεί δύο προβλήματα. Πρώτον, ότι ποτέ δεν υπήρχε πρόβλημα με την ε, περιοριστική δημοσιονομική πολιτική, ακόμη και όταν έπρεπε εσείς να την επιβάλλετε, παραβιάζοντας την εντολή σας για λόγους ε, συγκράτησης του πληθωρισμού. Και μιλάμε για μεγάλες περιόδου την τελευταία δεκαετία. Και το δεύτερο πρόβλημα που προκαλείται είναι ότι καταλήγουμε στο συμπεράσμα ότι η νομισματική πολιτική μεμονωμένα δεν είναι στην ουσία ε, μέρος της εντολής της ΕΚΤ. Όμως τα προηγούμενα χρόνια και σε μεγάλα διαστήματα είδαμε ότι παρά τις προσπάθειες ε, δεν κατάφερε να εξηγιάνει αυτά που είχε αναλάβει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρόλα αυτά παραβιάζοντας την εντολή της. Και η δεύτερη ερώτησή μου έχει να κάνει με την ε, οικονομική, χρηματοοικονομική σώρευση. Η ΕΚΤ ασχολείται πολύ με τον κατακαιρματισμό του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αυτό ισχύει και στην Πορτογαλία ε, και σας απασχολεί πώς θα προωθήσετε την συγκέντρωση σε τραπεζικό επίπεδο. Αυτό το θέμα πώς το βλέπετε, διότι μου φαίνεται ότι από αυτήν την έννοια οι ανησυχίες αυτές της ΕΚΤ έχουν σχέση και με λύσεις που έχουν βρεθεί για το χρηματοπιστωτική κρίση, ιδίως για τη διάσταση των τραπεζών και αυτά τα μέτρα που είχαν βρεθεί εκεί. Yes. Ευχαριστώ για τις τόσο ενδιαφέρουσες ερωτήσεις σας. Με τη σειρά. Για την ε, αναθεώρηση της στρατηγικής μας. Νομίζω ότι χτες η κυρία Λαγκάρτ διευκρίνησε ότι η αναθεώρηση θα λάβει χώρα συνολικά και με ανοιχτό πνεύμα και θα λάβει υπόψη όλα τα στοιχεία της νομισματικής πολιτικής σε ποιο περιβάλλον ασκείται η νομισματική πολιτική, ποια είναι η οικονομική κατάσταση διεθνώς, ποιο είναι το δημοσιονομικό επίσης ε, τοπίο και όλα αυτά θα ε, εξεταστούν κατά την αναθεώρηση της ε, στρατηγικής μας. Τώρα δεν ξέρω πόσο συνολική θα μπορούσε να είναι αυτή η αναθεώρηση, αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσε να πάει αρκετά μακριά ώστε να εξετάσει και το τι μπορεί να κάνει η δημοσιονομική πολιτική, η οποία σαφώς και βρίσκεται εκτός αρμοδιοτήτων της ΕΚΤ. Είναι οι αιρετοί οι οποίοι αποφασίζουν για την πολιτική αυτή. Τώρα λέτε ότι κατά το παρελθόν η ΕΚΤ ζητούσε περιοριστικές πολιτικές. Νομίζω ότι ο πρόεδρος Ντράγκη αλλά και η πρόεδρος Λαγκάρντα όποτε χρειάστηκε είπαν και έγινε και πολύ πρόσφατα, ε, μίλησαν για διαφορετικές πολιτικές, για επεκτατική δημοσιονομική πολιτική για παράδειγμα. Ε, ζήτησαν από τις χώρες που έχουν κάποιο δημοσιονομικό περιθώριο, κάποιο πλεόνασμα να το χρησιμοποιήσουν για να βοηθήσουν την σταθερότητα τιμών και άρα χρειάζεται όθηση στην ε, εσωτερική ζήτηση. Να χρησιμοποιηθεί σαν μοχλός δηλαδή η δημοσιονομική πολιτική. Οπότε η ΕΚΤΕ όντω έχει ζητήσει πολλές και διάφορες πολιτικές και κάποια στιγμή για κάποιο λόγο ζήτησε δημοσιονομικές πολιτικές και τώρα επίσης ζητάει επεκτατικές πολιτικές από τις χώρες εκείνες οι οποίες έχουν κάποιο δημοσιονομικό περιθώριο και ζητάει από άλλες χώρες μέλη που δεν έχουν αυτό το περιθώριο να ξαναδούν τη σύνθεση των ε, δαπανών τους ώστε να είναι πιο φιλικές προς την ε, οικονομική μεγέθυνση. Εγώ δεν είμαι προκατελημένος, όχι, είμαι υπέρ της σταθερότητας των τιμών Πού είναι και η αρμοδιότητά μας. Στη δημόσια συζήτηση που γίνεται από την ΕΚΤ με τον κόσμο, όλα συζητιούνται. Τώρα, για το δεύτερο, υπάρχουν εδώ πέρα ο κατακαιρματισμός. Έτσι, υπάρχουν δύο στοιχεία. Υπάρχει κατακαιρματισμός στην ίδια την Ευρωζώνη. Και είναι κάτι που δεν θα πρέπει να έχουμε. Είναι ο κατακαιρματισμός, κάτι που εμποδίζει την ε, ήπια λειτουργία και την απρόσκοπτη της νομισματικής πολιτικής. Ενώ τώρα αυτό δεν γίνεται. Η ΕΚΤ προσπαθεί να αποφύγει τον κατακαιρματισμό της νομισματικής και τραπεζικής αγοράς στην Ευρωζώνη. Και έχουμε δει τι απέδωσαν οι πολιτικές αυτές με τα επιτόκια καταθέσεων, το ρίμπορ, τις ε, δευτερογενείς αγορές. Όλα αυτά έδειξαν ότι ο κατακαιρματισμός που αυξήθηκε μετά την οικονομική κρίση μειώθηκε τώρα. Και τώρα η ΕΚΤΑ βοηθάει ολόκληρη την ε, Ευρωζώνη. Το too big to fail είναι ένα θέμα βέβαια. Είναι θέμα εποπτείας και εξυγένσης. Οι κανόνες οι σχετικοί εισήχθηκαν για να αντιμετωπιστεί το θέμα το too big to fail. Και η φιλοσοφία μας τώρα είναι ότι δεν υπάρχει κανονικά τράπεζα που να είναι too big to fail. Και αυτή βέβαια είναι η πρόκληση για το πώς θα γίνει η εξυγίανση, η οποία εξυγίανση ακριβώς αυτό το σκοπό έχει να αντιμετωπίσει το too big to fail. Συνεπώς, δεν είχαμε μέχρι τώρα βοήθεια. Υπάρχει το πρόβλημα ακόμα, είναι αλήθεια. Πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου προσπαθεί ακριβώς να το αντιμετωπίσει. Ευχαριστούμε. Ματουσέλο Ελκ. Ευχαριστώ για τα σχόλια που έκαναν ήδη οι συνάδελφοί μου, εν μέρει καλύφθηκα για την πρόταση που λάβαμε εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Ε, προφανώς πάντοτε υπήρξε η Τράπεζα της Ιταλίας, η της ένα φυτόριο για τα μεγάλα ταλέντα της χώρας μας. Και ξέρουμε πολύ καλά πόσο πλούσιο είναι το βιογραφικό του κυρίου Πανέτα. Μία ερώτηση λοιπόν εδώ υπάρχει κάποιο, δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα το οποίο να μας ενθουσιάζει μέχρι δακρύων. Ε, ξέρουμε τι γίνεται με το επίπεδο 3 και τις διάφορες στηρίδες που προλεγούνται γι' αυτό στην Ιταλία, τη Γερμανία και την Αυστρία. Η Ιταλία ιδίω θα πληγεί περισσότερο από αυτό το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί. Χωρί να μπούμε στι λεπτομέρειε ε, του μηχανικού αυτού προγράμματο που ανακοινώνεται σήμερα, θεωρείται ότι το μέλλον των τραπεζών θα είναι πάντοτε περισσότερο προ την κατεύθυνση των ψηφιακών υπηρεσιών και θα χάνονται θέσει εργασία. Και κυρίω τι μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε επί τη ουσία να υπάρξει απερίμωση στην απασχόληση στον κλάδο αυτό. Well, thank, thank you, Ευχαριστώ κύριε Μαρτουσέλο. Βεβαίως, να μην σχολιάσω το τι γίνεται με τους μεμονωμένους διαμεσολαβητές και το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε χθες είναι ένα πράγμα. Από την άλλη, θα πρέπει να υπάρξει κάποια αναδιάρθρωση στις τράπεζες βάσει των τεχνολογικών, λόγω μάλλον, των τεχνολογικών εξελίξεων που πλήττουν και τον τραπεζικό τομέα. Θα, του έλεγα, θα τους έλεγα τεχνολογικούς κραδασμούς. Βεβαίω τώρα για την ΕΚΤ, επειδή εμεί είμαστε το, η κεντρική έδρα των τραπεζικών εξελίξεων, πρέπει να πω ότι εμεί τουλάχιστον βρισκόμαστε σε μετάβαση σε μετάβαση από τον παραδοσιακό τρόπο λειτουργία μα ε, για την ε, εμπορική λειτουργία μιας τράπεζας, στην νέα οργάνωση της τράπεζας μετά το κύμα των τεχνολογικών εξελίξεων που αναδύεται τώρα. Και όπως είχα πει και προηγουμένως, οι τράπεζες αντιμετωπίζουν τώρα έναν πολύ στιγνό ανταγωνισμό από εξωτραπεζικούς ε, φορείς. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι την ερχόμενη πενταετία, δεκαετία, 60% των εισοδημάτων της λιανικής λειτουργίας των τραπεζών θα έχει απειληθεί και κλαπεί από τις εταιρείες FinTech. Το χρηματοπιστωτικό λοιπόν το οποίο διαμορφώνεται εντελώ διαφορετικά. Οι τράπεζε θα πρέπει να αναθεωρήσουν τη σχέση κεφαλαίου προσωπικού, μειώνοντα το προσωπικό, αυξάνοντα το κατά πόσον χρησιμοποιώντα τεχνολογικού πόρου και βεβαίω αυτό αλλάζει πολύ το πώ λειτουργούν οι τράπεζε αλλά και τι προσφέρουν στο κοινό. Θα προσφέρουν καλύτερε υπηρεσίε σε χαμηλότερο κόστο και με τρόπο ασφαλέστερο. Βεβαίω, θα υπάρχει κοινωνικό κόστο. Αυτό είναι πάντα το τίμημα όταν βρίσκεται κάποιο σε μετάβαση από τον ένα τομέα στον άλλο. Είμαστε τώρα ακριβώ σε αυτή τη φάση. Σε πολλές χώρες, ε, μεταξύ των οποίων και η Ιταλία, οι τράπεζες έχουν μια είδους αντασφάλιση. Δηλαδή, κοιτάζουν να προσφέρουν ποσά στην διευκόλυνση της μετάβασης αυτής. Αυτό γίνεται και στην Ιταλία και σε άλλε χώρε τη Ευρωζώνη και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Αλλά δεν μπορούμε να ανακόψουμε το τεχνολογικό κύμα. Διότι θα έχουμε ένα σύστημα πολύ αποδοτικότερο με φτηνότερε υπηρεσίε, με αποτελεσματικότερε υπηρεσίε στην πραγματική οικονομία εν γέννη. Σε ιδιώτε, σε εταιρείε και ιδίω στι μικρέ εταιρείε. Διότι ω τώρα περισσότεροι, τα περισσότερα από τα πάγια και το πρόβλημα, το, το κόστος του τραπεζικού τομέα βαρύνει τις μικρότερες επιχειρήσεις και εταιρείε. Έτσι θα αλλάξουν και οι συνθήκες χρηματοδότησής τους αυτές των μικρομεσαίων και αυτό βεβαίως είναι μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τελευταία ερώτηση. Εύελιν Ρέγνερ, Σοσιαλδημοκράτης. Ευχαριστώ πολύ. 2019 έχουμε, γερμανικά μιλάω. 2019 έχουμε λοιπόν. Και κοιτώντας την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, και το Διοικητικό Συμβούλιο, βλέπουμε ότι απέχουν πολύ όσον αφορά τη συμμετοχή ανδρών και γυναικών. Τέσσερις άντρες, δύο γυναίκες. Ε, και η γυναίκα που διορίστηκε διαδέχεται η γυναίκα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, έχει επανειλημμένα πει ότι δεν μπορεί να συνεχίσετε έτσι. Εσείς ε, είπατε κάτι πολύ ενδιαφέρον στην εισήγησή σας. Μήπως μπορείτε να το αναπτύξετε περαιτέρω. Πώς θα πρέπει να πετύχουμε όσο γίνεται πιο διαφοροποιημένη συμμετοχή, τι θα πρέπει να γίνει σε επίπεδο ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εσεί εσείς αναφερθήκατε στο παράδειγμα της ε, Ιταλικής Τράπεζας. Ε, εσείς πώς πιστεύετε ότι μπορεί να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στην εισήγησή μου και στις απαντήσεις μου προσπάθησα να σας περιγράψω τι έκανα και τι μπορώ να κάνω ως ε, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Κεντρικής Τράπεζας, ε, διότι τώρα είμαι μέλος της, ε, του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ιταλίας. Έχω λάβει υπόψη μου την ανάγκη για διαφοροποίηση στην Κεντρική Τράπεζα σε πολλούς τομείς και όσον αφορά την ισορροπία των δύο φύλων. Προσπάθησα λοιπόν να σας δώσω μια εικόνα του τι μέτρα μπορεί να λάβει ένας φορέας, ένας οργανισμός για καλύτερη ισορροπία των δύο φύλων. Και σας έδωσα το παράδειγμα της Τράπεζας της Ιταλίας, όχι επειδή θεωρώ ότι είναι πιο ε, σημαντικό από άλλα, αλλά σε αυτό συμμετείχα. Συμμετείχα στη διοίκηση πολύπλοκου οργανισμού με 8.000 υπαλλήλους, όπου είχαμε πολύ κακή, ε, δεν είχαμε καθόλου ισορροπία ανάμεσα στα δύο φύλλα. Αυτό το συνειδητοποίησα όταν ανέλαβα ε, καθήκοντα. Δεν μας άρεσε αυτό και προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Σας ε, παρουσίασα λοιπόν τα αποτελέσματα που έχουμε πετύχει μέχρι τώρα, τα χρόνια δηλαδή που ήμουν εγώ στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και φυσικά θα κάνω το ίδιο εάν και εφόσον ε, διοριστώ στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής ε, του Διοικητικού Συμβουλίου, συγγνώμη, ε, δεν είναι κάτι στο οποίο μπορώ να επέμβω. Δεν έχω καμία δυνατότητα να ασκήσω επιρροή στα κράτη-μέλη. Νομίζω όμως ότι είναι προς συμφέρον όλων να έχουμε ισορροπημένη σύνθεση σε κάθε συμβούλιο όσον αφορά τα δύο φύλλα. Αλλά φυσικά δεν μπορώ να αναλάβω δεσμεύσει στο όνομα ε, του Διοικητικού Συμβουλίου ή των άλλων μελών του, της Εκτελεστικής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ τον ε, κύριο Πανέτα. Λίγη εδώ η ε, ακρόαση και μπορούμε να συνεχίσουμε. Δύο λεπτάκια διάλειμμα για να επιτρέψουμε στην επόμενη υποψήφια να εισέλθει στην αίθουσα. Okay, thank you very much. I... Ευχαριστούμε πολύ. Ας ξεκινήσουμε. Τώρα λοιπόν χαίρομαι που υποδέχομαι εδώ την Ιζαμπέλ Σνάμπελ που είναι υποψήφια για τη θέση Τη Εκτελεστική επιτροπή τη Ευρωπαϊκή Κυριακή Τράπεζα. Στι 25 Σεπτεμβρίου η Σαμπίν Λόντον Σλάγερ, που είναι μέλο ακριβώ Εκτελεστική επιτροπή, ενημέρωσε τον πρόεδρο Τράγκη ότι 31 Οκτωβρίου 2019 παρετείται πριν από τη λήξη τη θητείας τη. Σύμφωνα με το άρθρο 283.2 τη συνθήκη για την Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωμοδοτεί μετά από σύσταση του Συμβουλίου για τον ορισμό μέλους της ε, Εκτελεστικής Επιτροπής. Έτσι λοιπόν υπήρξε ε, συνομιλία του Συμβουλίου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κάλυψη της θέσης Εκτελεστικής Επιτροπής για 8 χρόνια από 1η Ιανουαρίου του 2020. Πριν από τη σημερινή ακρόαση στείλαμε στην υποψήφια ερωτήσεις, 55 ερωτήσεις και οι απαντήσεις της υποψηφίας επισυνάπτονται στην έκθεση της σύστασης του Συμβουλίου. Επίσης, μετά την ακρόαση θα ακολουθήσει ψηφοφορία στις 5 το απόγευμα σήμερα το απόγευμα. Η Επιτροπή ΕΚΟΝ θα υποβάλει πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, για απόφαση βάσει της σύστασης του Συμβουλίου όσον αφορά τον ορισμό της στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ. ψηφοφορία θα γίνει στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου, 16 με 19 Δεκεμβρίου. Στην αρχή της ακρόασης θα ακούσουμε μια σύντομη εισαγωγή 10 λεπτών από την υποψήφια και θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και απαντήσεις. Συνεπώς, κύριε Σνάβελ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Αξιότιμη πρόεδρος, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, με τιμή και ταπεινότητα αντιμετωπίζω την υποψιότητά μου ως μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εκτιμώ όλους ιδιαίτερο τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή ορισμού. Αποτελεί μέρος της λογοδοσίας της ΕΚΤΕ που είναι ένα αναγκαίο αντίβαρο στην ανεξαρτησία της και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω την ευκαιρία να ανταλλάξω απόψεις μαζί σα και στη συνέχεια να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Στις αγωγικέ μου παρατηρήσεις θα ήθελα να συζητήσω την νομισματική πολιτική της ΕΚΤ και τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Ευθύς εξ αρχή θα σας πω όμω κάποια λόγια για τα δικά μου προσόντα η επαγγελματική μου σταδιοδρομία. Ήμουνα ερευνήτρια και σύμβουλο πολιτική σε θέματα νομισματικά και οικονομικά. Έχω συγκεντρώσει εμπειρία σε θέματα συμβουλών πολιτική, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχω δει πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχει κανεί στην ε, δημόσια συζήτηση και να επικοινωνεί με αποτελεσματικό τρόπο. Ως ερευνήτρια λοιπόν έχω μελετήσει οικονομικές κρίσεις, οικονομικούς ε, κανόνες ε, και ροές κεφαλαίων διεθνώς για πάρα πολλά χρόνια. Και η έρευνά μου είχε να κάνει με το too big to fail, τα θέματα αυτά που αντιμετώπισε το γερμανικό τραπεζικό σύστημα στην ε, κρίση του 1939. Έπειτα διαπίστωσε ότι για 400 χρόνια οι φούσκες των τιμών έχουν οδηγήσει σε κρίσεις, όπως επίσης και το ξεπούλημα, ε, πολύ φθηνές πωλήσει δηλαδή, και κάθισα να σκεφτώ τι μπορούν να κάνουν οι κεντρικές τράπεζες. Και είπα τι είναι αυτό που καταστρέφει τελικά την οικονομική ολοκλήρωση και τι ήταν αυτό που οδήγησε στην τελευταία κρίση. Και ο Σύμβουλο Πολιτική συνεισέφερα στη συζήτηση τόσο στη Γερμανία όσο και στην Ευρώπη για οικονομικά ζητήματα. Συμμετέχω στο Γερμανικό Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων που συμβουλεύει τη γερμανική κυβέρνηση και το ευρύτερο κοινό, όντα όμω πλήρω ανεξάρτητο όργανο. Και είμαι αντιπρόεδρο τη Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου και έχω συμμετέχει και στις συζητήσεις για την οικονομική σταθερότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είμαι και συμπρόεδρος του Γαλλογερμανικού γερμανικου Συμβουλίου ε, Οικονομολόγων Εμπειρογνωμόνων που δημιουργήθηκε βάσει τη συμφωνία του Άχεν από τη Γαλλική και τη Γερμανική κυβέρνηση. Όλες αυτές οι δραστηριότητε μου ε, οδηγούν στο να προσπαθήσω να αντιμετωπίσω το θέμα από διαφορετικές οπτικές γωνίες και να συμβάσω όλες αυτές τις ε, οπτικές γωνίες σε μια συνεπή πολιτική πρόταση. Έχω εκτιμήσει τις συζητήσεις που έχω κάνει και τους διαλόγους μου με κάθε πλευρά, με πολιτικούς, με επαγγελματίε και το κοινό γενικά και χρησιμοποιώ τις γνώσεις μου αυτές και τις αρχές μου για να παρουσιάσω τις απόψεις μου και κάθε φορά που έδινα συνεντεύξεις ή έγραφα άρθρα εξηγώ τις περίπλοκες σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα σε όλα αυτά και αυτό με κατανοητό τρόπο. Τώρα έρχομαι στην νομισματική πολιτική της ΕΚΤΑ. Πρόσφατα χρόνια η Ευρωπαϊκή η Ευρωζώνη μάλλον αντιμετώπισε ε, προβλήματα ε, χαμηλής ανάπτυξης και μεγάλης ανεργίας. Οι έρευνες δείχνουν ότι η έκτη ενισέφερε σημαντικά στο να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Και τώρα έχουμε καταλήξει σε μια απειλή αποπληθωρισμού. Και εξαιτία επίση των εμπορικών συγκυριών και τη ανερχόμενη αβεβαιότητα, βλέπουμε μια επιβράδυνση της οικονομικής μεγένθησης που επηρεάζει την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη και κυρίως στη μεταποίηση. Σαν συνέπεια, ο πληθωρισμός προβλέπεται να παραμείνει πολύ χαμηλότερο από το στόχο μας, που είναι το κάτω, αλλά κοντά στο 2% και αυτό μεσοπρόθεσμα. Γι' αυτό το Σεπτέμβριο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε να επεκτείνει την νομισματική πολιτική ώστε να αντιμετωπιστούν αυτές οι εξελίξεις και να μπορέσει να τηρήσει την εντολή της που είναι σταθερότητα τιμών. Και επειδή υπάρχουν πιο αδύναμες πιέσεις επί το τιμών, οι αποφάσεις αυτές δικαιολογούνται. Όμω, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η νομισματική πολιτική τώρα αντιμετωπίζει σημαντικέ προκλήσει που πρέπει να αντιμετωπιστούν και αυτέ και επιπλέον και οι παρενέργειέ τη. Η εμπειρία των πρόσφατων ετών έχει δείξει ότι είμαστε σε χαμηλότερα επίπεδα από το μηδέν. Παρ' όλα αυτά μπορεί να υπάρχει και ένα όριο που να είναι λιγότερο αποτελεσματική νομισματική μας πολιτική και αυτό είναι που ονομάζουμε reversal rate, δηλαδή όριο πέρα από το οποίο αντιστρέφεται η θετική επίδραση των μέτρων. το τόνισε και η κυρία Λαγκάρντα ότι μπορούμε να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο και να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής. Άρα να χρησιμοποιήσουμε το δημοσιονομικό χώρο εκεί όπου αυτός υπάρχει και να έχουμε μια ε, καλύτερη και πιο αποτελεσματική, πιο φιλική προς την ανάπτυξη σύνθεση των δημοσίων δαπανών. Επιπλέον υπάρχουν και ανησυχίες για τις ε, παρενέργειες. Ε, αυτές οι ανησυχίες πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη, γιατί αν υπάρξουν τέτοια φαινόμενα μπορεί να αποδυναμώσουν την οικονομία και να απειλήσουν τη σταθερότητα τιμών. Είδαμε ότι επειδή έχουμε χαμηλά επιτόκια, οι επενδυτές προσπαθούν να βρουν άλλες επενδύσεις υψηλότερων αποδόσεων ε, όπως επίσης το αποτέλεσμα των υψηλών τιμών ενεργητικού και η χαμηλή αποζημίωση σε αυτόν που παίρνει ρίσκο επίσης αποσταθεροποιούν την κατάσταση. Τέτοιες ε, εύθραυστες καταστάσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται με μακροπροληπτικές πολιτικές που μπορούν βέβαια να ε, διορθωθούν ανάλογα με την κατάσταση της ε, κάστοτε αγοράς ή χώρας. Προσπαθούμε να βρούμε το καταλληλότερο χρόνο για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αυτές, να είμαστε πιο ανθεκτικοί και να αντιμετωπιστούν και οι αντικυκλικές ε, επιδράσεις. Και αυτό με διάφορα μακροπροληπτικά ε, εργαλεία και επίσης μπορούν και οι μη τράπεζες να αναπτυχθούν αντίστοιχα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει να παίξει σημαντικό ρόλο. Τώρα, πέρα από τι επιπτώσει του οικονομικού συστήματο, πολλοί ε, πολίτε ανησυχούν ε, για τα χαμηλά επιτόκια και το πώ αυτά επιδράζουν την καθημερινότητά του. Ανησυχούν για τι αποταμιεύσει του και τι συντάξει του και ανησυχούν ότι θα αντιμετωπίσουν αρνητικά επιτόκια στι αποταμιεύσει του. Η ΕΚΤ πρέπει να ακούει πάρα πολύ προσεκτικά αυτέ τι ανησυχίε. Η πρόεδρο έχει ήδη πει ότι η ΕΚΤ θα προχωρήσει σε μια συνολική αναθεώρηση του πλαισίου τη νομισματική πολιτική. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να συμπεριλάβει και την ανάλυση των παρενεργειών που μπορεί να επηρεάζουν τη μετακύληση της νομοθετικής πολιτικής. Επιπλέον ανακοίνωσε ότι η επικοινωνία με το κοινό θα αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΚΤ. Και εγώ πολύ θα χαρώ να αποτελέσω μέρο τη προσπάθεια αυτή. Να εξηγήσω τη λογική και τι επιπτώσει τη νομισματική πολιτική τη ΕΚΤ είναι κάτι πολύ βασικό για να διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στην κεντρική του τράπεζα. Συγχρόνω πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τα χαμηλά επιτόκια στην Ευρωζώνη δεν είναι μόνο θέμα τη ΕΚΤ. Γιατί οι μακροπρόθεσμε εξελίξει στα επιτόκια που έχουν να κάνουν και με διαρθρωτικέ αλλαγέ, με τη δημογραφική αλλαγή, αλλαγή, την αλλαγή στην παραγωγικότητα. Οπότε όλα αυτά επηρεάζουν την κατάσταση. Επιπλέον απαιτούν και οικονομικές πολιτικές που να προσανατολίζονται στο μέλλον και να στηρίζονται στην παραγωγικότητα και την καινοτομία. Η νομισματική πολιτική μπορεί να στηρίξει, αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει οικονομικές πολιτικές υπέρ της ανάπτυξης. Και γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε στόχους φιλόδοξης πολιτικής υπέρ της καινοτομίας και των επενδύσεων με ενέργεια, εκπαίδευση, και ψηφιακέ αλλά και μη ψηφιακέ υποδομέ. Επιπλέον, για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση χρειάζεται ε, μια πραγματική ε, ευρωπαϊκή τραπεζική και κεφαλαϊκή αγορά που να αντιμετωπίζει τα σόκο, να προστατεύει τα νοικοκυριά, τι αποταμιεύσει και να προτείνει μέτρα που να είναι ικανοποιητικά για όλους πρέπει να συμπληρωθεί η Τραπεζική Ένωση, η Κεφαλιακή Επίση Ένωση, για να υπάρχει ολοκλήρωση των αγορών και να μειώνονται κίνδυνοι. Επιπλέον, μία ευρωζώνη με αντοχή θα δημιουργήσει ένα δημοσιονομικό πλαίσιο που θα επιτρέπει στις ε, αντικυκλικές ε, πολιτικές να προωθούν τις επενδύσεις αλλά να έχουν και δημοσιονομική σταθερότητα. Οι συστάσεις, ε, οι γερμανικές και οι γαλλικές, η έκθεση που ονομάζεται 7 συν 7 έχει συνεισφέρει σε αυτό και συμπεριλαμβάνει ένα βασικό μήνυμα. Σταθεροποίηση της Ευρωζώνης απαιτεί μια ισορροπημένη προσέγγιση κινδύνων και πειθαρχία στην αγορά που να συμπληρώνουν το ένα το άλλο. Και ενώ η πειθαρχία χρειάζεται για να υπάρχουν καλά κίνητρα, ο πλημμυρισμό του κινδύνου σταθεροποιεί την οικονομία και αποφεύγει συστημικέ κρίσει. Πρέπει να συμπληρωθεί η Οικονομική και Ένωση. Η οικονομική πολιτική πρέπει να ασχοληθεί όμω και με την κλιματική αλλαγή, που αποτελεί την πιο σημαντική πρόκληση του 21ου αιώνα. Οι κεντρικέ τράπεζε φυσικά και έχουν να παίξουν ένα ρόλο και να διασφαλίσουν ότι εξακολουθούν να τηρούν την εντολή τους. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, αυτό είναι που θα δούμε στην αναθεώρηση της νομισματικής πολιτικής. Επιπλέον, η ψηφιακή τροποποίηση έχει αλλάξει και την εποπτεία αλλά και τη λειτουργία των τραπεζών. Η ΕΚΤΕ πρέπει να εξετάσει τις επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στις πολιτικές της, χρησιμοποιώντας βέβαια και τις ευκαιρίες που αυτές προσφέρουν. Και καταλήγω. Το πρόσφατο ευρωβαρόμετρο έδειξε ότι η εμπιστοσύνη στο ευρώ βρίσκεται στα υψηλότερα ποτέ από την αρχή που το ερευνάμε το θέμα. Και η έχει συνεισφέρει πολύ σημαντικά σε αυτές τις θετικές εξελίξεις. Έχει αποδειχτεί ότι είναι ένα αποτελεσματικό όργανο που τηρεί την εντολή του διασφάλιση σταθερότητας τιμών. Εάν επιβεβαιωθώ στη θέση μου, θα είμαι περήφανη να αποτελέσω μέρο του οργάνου αυτού Εφόσον επιβεβαιωθώ στη θέση αυτή, θα συνεισφέρω με όλη μου την ενέργεια στη διαμόρφωση πολιτικής της έκτα επόμενα 8 χρόνια και να τονίσω 8 χρόνια προς όφελος ολόκληρης της Ευρωζώνης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και τώρα περιμένω τι ερωτήσεις σας και προσβλέπω στη συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στις ερωτήσεις. Ξεκινάμε με τον Μάρκους Φέρμπερ από το ΕΛΚΑ. Σας ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπετε θα μιλήσω τη μητρική μας. Σας καλωσορίζω και χαίρομαι που για δεύτερη φορά η πατρίδα μου έχει προτείνει γυναίκα. Ε, αυτό ας είναι παράδειγμα για άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χαίρομαι που Είπατε ότι θέλετε ε, να σπάσετε την παράδοση που υπάρχει όσον αφορά τους άλλους ε, Γερμανούς προκατόχους σας ε, και να παραμείνετε στη θέση επί 8 χρόνια όσον αφορά την ε, τελευταία δέσμη μέτρων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είπατε στην ε, Handelsblatt ότι δεν ε, είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο, δεν μας απειλεί κάποιο σπιράλ προς τον πάτο και στις γραπτές σας ε, απαντήσεις ε, υπαριθμών 5 ε, υπερασπιστήκατε τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ποια κυρία Σνάμπελ να πιστέψω, αυτήν που έδωσε συνέντευξη στις 15 Ενάτου στη Χάντελσπλατ ή το ή αυτά που ακούω τώρα, τι θα κάνετε όταν αναλάβετε καθήκοντα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Φέρμπερ. Συγχωρήστε με, θα απαντήσω στα αγγλικά. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα και σημαντική αυτή ερώτηση. Όπως είπα κατά την εισήγησή μου, οι αποφάσεις του Σεπτεμβρίου αντικατοπτρίζουν την παγκόσμια επιβράδυνση της οικονομίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο ε, η εμπορική διαμάχη έχει οδηγήσει σε επιβράδυνση στο παγκόσμιο εμπόριο, την παγκόσμια ανάπτυξη και αυτό φαίνεται και στην Ευρωζώνη. Οι προβλέψεις για την ανάπτυξη έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω και ε, οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό είναι πιο αρνητικές από ό,τι ήταν πριν. Γι' αυτό ήταν σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έπρεπε να αναλάβει δράση και να εφαρμόσει επιπλέον μέτρα για να αντισταθμίσει αυτές τις αρνητικές εξελίξεις. Ε, αλλά τίθεται το ερώτημα τι θα πρέπει να γίνει. Το Διοικητικό Συμβούλιο συμφώνησε και εγώ θα συμφωνούσα ότι χρειαζόταν ε, μια σαφής θέση και συζητήθηκε το ποια μέσα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Συζητήθηκε, για παράδειγμα, να μειωθεί το επιτόκιο στη διευκόλυνση των καταθέσεων. Ε, συμφωνήθηκε... Έγινε συμφωνία όσον αφορά ε, τις ε, στοχευμένες μακροπρόθεσμες επιχειρήσεις πράξεις αναχρηματοδότησης, αλλά στο στη συνέντευξή μου ε, ε, προσπαθούσα να πω ότι εγώ μάλλον θα περίμενα όσον αφορά την αγορά στοιχείων του ενεργητικού. Δεν νομίζω ότι ήταν απαραίτητο να ξεκινήσει ήδη τότε αυτό. Θα ήθελα να τονίσω όμως ότι αυτό μπορεί παρόλα αυτά να δικαιολογηθεί εντό τη εντολή τη Ευρωπαϊκής Κεντρικής τράπεζα και η συζήτηση σχετικά με το αν θα πρέπει να ξεκινήσει η αγορά στοιχείων του ενεργητικού ξεκίνησε τελικά υπήρξε πλειοψηφία ότι θα πρέπει να ξεκινήσει πάλι η αγορά. Και ε, των διαδικασιών λήψης αποφάσεως αυτό ήταν πια η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Εγώ αν ψήφιζα ίσως ε, να ε, είχα ψηφίσει να περιμένουμε. Αλλά τελικά μάλλον η απόφαση θα ήταν η ίδια που ήταν και τώρα. Η στάση όσον αφορά την νομισματική πολιτική είναι όντως ε, πολύ προσαρμοστική. Ελπίζουμε λοιπόν ότι αυτό θα αρκέσει ώστε να επανέλθει ο πληθωρισμός στον στόχο του κοντά αλλά μόλις κάτω από το 2%. Θα πρέπει να δούμε τι θα συμβεί. Όλα αυτά εξαρτώνται από το τι θα συμβεί και στην οικονομία. Αυτή τη στιγμή τα δεδομένα δεν ήταν τόσο αρνητικά όσο ε, υπήρχε φόβος. Η Γερμανία, για παράδειγμα, δεν μπήκε σε τεχνική ύφεση, παρότι ε, πολλοί το είχαν προβλέψει αυτό. Ήταν λοιπόν κάπως πιο ευνοϊκές εξελίξεις από ό,τι φοβόμασταν. Ε, Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να είμαστε ε, αισιόδοξοι ότι δεν θα περάσει σε ύφεση η ζώνη του ευρώ και γι' αυτό είμαι και αισιόδοξη ότι μέσω πρόθεσμα ο πληθωρισμός θα κινηθεί προς τον στόχο παρότι μάθαμε ότι αυτό μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από ό,τι περιμέναμε αρχικά. Σας ευχαριστώ πολύ, ο Άλφρετ Σαντ από το S&D. Σας ευχαριστώ στις απαντήσεις σας πριν τη σημερινή συνεδρίαση. Αναφερθήκατε επανειλημμένα στις διαφορετικές αλλαγέ. αναφερθήκατε στην έλευση των κρυπτονομισμάτων, την καταπολέμηση του ξεπλήματο χρήματο, την δημογραφική αλλαγή και ε, τις ε, των υποδομών. Αναφερθήκατε και στην ανάγκη να ε, ρυθμίσουμε τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μα για να αντιμετωπίσουμε αυτέ τι προκλήσει. Ε, σύμφωνα με τους κανόνες όμως ε, Όσον αφορά τον πληθωρισμό και το δημόσιο χρέος, βρισκόμαστε κοντά στην κατάσταση που βρισκόμαστε ε, τη ε, δεκαετία του 1990 και ε, το θέμα είναι αν συνεχίζουν να είναι εύστοχα τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν τότε σήμερα. Νομίζω ότι θα πρέπει να διασκεδαστούν αυτές οι αμφιβολίες αν θέλουμε να αποφύγουμε διαταράξεις στα οικονομικά μα συστήματα. Θα πρέπει να έχουμε τα εργαλεία για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να συμμετέχει σε μια αξιολόγηση τέτοιων νέων μέσων και αν ναι, πώς. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση αυτή. Ε, αυτό είναι πολύ μεγάλο ερώτημα, οι διαρθρωτικές αλλαγές, ε, τι αλλαγές επιφέρουν στην οικονομία μας. Ε, όπως είπατε, έχουμε δει τεράστιες διαρθρωτικές αλλαγές, δημογραφική αλλαγή, ψηφιακή επανάσταση. Έχουμε και την αλλαγή του κλίματος και είναι σαφές ότι αυτό θα αλλάξει πολλά πράγματα στην οικονομία μας και αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται και στην οικονομική πολιτική. Φυσικά θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι πολλές από τις αλλαγές αυτές ε, πραγματοποιούνται εδώ και πολύ καιρό. Δεν ε, έχουμε κάτι ανατρεπτικό εδώ πέρα από την ε, οικονομική κρίση, αλλά όλες οι άλλες προκλήσεις που περιγράφεται είναι κάτι που συμβαίνει εδώ και πολύ καιρό. Και γενικά νομίζω ότι οι οικονομίες μας έχουν ε, καταφέρει να αντιμετωπίσουν αρκετά καλά αυτές τις αλλαγές, προσαρμόζοντας συνεχώς την πολιτική. Δεν νομίζω λοιπόν ότι χρειάζεται να αλλάξουμε το συνολικό σχεδιασμό της οικονομικής μας πολιτικής. Νομίζω ότι μας εξυπηρετεί ακόμα πολύ καλά, αλλά θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί απέναντι στις νέες εξελίξεις και να κάνουμε αλλαγές όπου αυτό φαίνεται απαραίτητο. Όσον αφορά λοιπόν την Κεντρική Τράπεζα, είναι σαφές ότι ένα σημαντικό θέμα είναι τα ψηφιακά νομίσματα. Όσον αφορά τα συστήματα πληρωμών, αυτά άπτονται και της νομισματικής πολιτικής. Βλέπουμε εδώ και αρκετό καιρό την ανάπτυξη κρυπτονομισμάτων. Ε, αρχικά αυτά ήταν νομι... δεν ήτανε... ήτανε νομίσματα, αλλά ήταν πιο πολύ ε, ε, εργαλεία κερδοσκοπίας. Δεν ε, εξυπηρετούσαν το ρόλο ενός νομίσματος, σπάνια χρησιμοποιούνταν ε, για πληρωμές. Τώρα όμως νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε νέα φάση με την πρόταση Λίμπρα που είναι διαφορετική, διότι η σημαντική διαφορά είναι ότι είναι σταθερό νόμισμα το οποίο ε, υποστηρίζεται από εγγύησεις. Έτσι η αξία του είναι πιο σταθερή και Ε, η ιδέα αυτή συνδέεται με το τεράστιο δίκτυο του Facebook που δίνει σε αυτό το νόμισμα τη δυνατότητα να γίνει παγκόσμιο νόμισμα. Και γι' αυτό όλοι ε, όσοι διαμορφώνουν την πολιτική θα πρέπει να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις τους τελευταίους μήνες συζητήθηκαν ε, εντατικά οι κίνδυνοι από τέτοια νομίσματα. Υπάρχουν κίνδυνοι για τους καταναλωτές που σχετίζονται με την προστασία του καταναλωτή. Υπάρχουν κίνδυνοι όσον αφορά τις παράνομες πληρωμές, ε, την νομοποίηση παράνομων εσόδων, ε, την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Ε, πράγματα που διευκολύνονται με τέτοια νομίσματα. Υπάρχουν ε, κάποιοι κίνδυνοι για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα, κάτι που πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μα. Ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη μα τον συστημικό χαρακτήρα τέτοιων πληρωμών. Και τέλο, μπορεί να υπάρξουν επιπτώσει στην μεταφορά τη διάδοση της νομισματικής πολιτικής. Και αυτό θα επηρεάσει άμεσα τις κεντρικές τράπεζες και γι' αυτό θα πρέπει να το ε, εξετάσουν πολύ προσεκτικά. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες ε, ε, ελλείψεις, κάποιες ανεπάρκειες του ισχύοντος συστήματος, αλλιώς δεν θα υπήρχαν αυτά τα νομίσματα. Και νομίζω ότι θα πρέπει να ενεργήσουν προορατικά οι κεντρικές τράπεζες. Το εάν θα μπορούσε να είναι εξίσου καλό το σύστημα TIPS που συζήτησε χθε ε, η ε, Πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Λουί Καρικάνο από το Ρινιού. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε που ήρθατε σε αυτή την επιτροπή. Πολλοί οικονομολόγοι ανέφεραν ε, στοιχεία σημαντικά για την οικονομία και διάφορα μελλοντικά σενάρια. Και εδώ έχουμε δει να συμβαίνει κάτι με το Brexit. Οι ψευδεί ειδήσει και οι λαϊκιστέ μετά από τρει δεκαετίε οδήγησαν το Ηνωμένο Βασίλειο να εγκαταλείψει την Ένωση. Κάτι παρόμοιο μπορεί να συμβεί και με την νομισματική πολιτική στο... στην Ευρωζώνη. Πολλά είναι τα κράτη που έχουν υποστεί πλήγματα νομισματικού εμ, λαϊκισμού με τσουνάμι ε, νομισματικά, με την... Ε, ηγεμονία κάποιων χωρών εναντί άλλων κτλ. Και πολλοί πολίτες πιστεύουν ότι μία τόν ετών απειλούνται λόγω της υιοθέτηση του ευρώ. Ε, στην Ευρωζώνη και ότι μπορεί να τις χάσουν. Τα επόμενα λοιπόν χρόνια και δεδομένου του κράτους προέλευσή σας, τα καθήκοντα που θα αναλάβετε δεν είναι πάρα πολύ απλά και δεν σας ζηλεύω. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει, κυρία Σνάμπελ, για να ξεπεράσουμε αυτά τα επικίνδυνα αφηγήματα. Θα προσπαθήσετε να προβάλλετε καλύτερα την πολιτική της έκτη για να καταλαβαίνει ο κόσμος καλύτερα και τι αποφάσει της ΕΚΤ. Τι έχετε υπόψη συγκεκριμένα. Και για να ολοκληρώσω να πω ότι ίσως να πιστεύετε ότι ο καθορισμός των επιτοκίων είναι η βασική σας δουλειά και θα είναι σίγουρα σημαντικό. Αλλά θα πρέπει να προβάλλετε σωστά και τη δουλειά της ΕΚΤ για να καταλαβαίνει ο κόσμος που χρησιμεύει μακροπρόθεσμα. Ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την πολύ χρήσιμη ερώτηση. Η ερώτηση αυτή με έχει απασχολήσει και δεν με έχει αφήσει να κοιμάμαι εδώ και καιρό. Λόγω των σχετικών συζητήσεων στη Γερμανία. Η συζήτηση στη Γερμανία πραγματικά με ανησυχεί όπως γίνεται, διότι έχουν πάρει επιθετικούς τόνους τα πράγματα και οι τοποθετήσεις. Η νομισματική πολιτική, και αυτό είναι το πρόβλημα, είναι πάρα πολύ περίπλοκη. Είναι πολύ λίγοι αυτοί που πραγματικά καταλαβαίνουν τι συμβαίνει. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ο κοινό πολίτη, το κοινό, να καταλαβαίνει τι κάνει η ΕΚΤ. Και είναι πολύ δύσκολο να χρησιμοποιηθεί ένα θεσμικό όργανο από, δι... από πομπαίου διότι κάποιο που απλώ ακούει αυτό το αφήγημα μπορεί να πιστέψει κατά 50% ότι είναι σωστό και 50% ότι είναι ψεύδος. Είναι πολύ δύσκολο να διακρίνει κανεί την αλήθεια. Συμφωνώ λοιπόν απολύτω. Πρέπει να ξεκινήσουμε με μια προσπάθεια ε, επιμορφωτική. Να εξηγήσουμε τι κάνει η νομισματική πολιτική σε πρώτη φάση. Βεβαίω αυτό έχει να κάνει και με τι γνώσει χρηματοοικονομικών. Κάτι που είναι μια πολύ ε, σημαντικότερη ευθύνη. Δεν μπορούν να την αναλάβουν οι κεντρικέ τράπεζε. Είναι δουλειά του εκπαιδευτικού συστήματος. Ε, εδώ πρέπει να κοιτάξουμε τα επιτόκια να μην γίνουν αρνητικά. Αλλά για τους οικονομολόγους αυτό που μετράει τα πραγματικά επιτόκια. Όμως 90% του πληθυσμού δεν καταλαβαίνει τη διάκριση των πραγματικών από τα αρνητικά επιτόκια. Οπότε πρέπει να κάνουμε μια σοβαρή προσπάθεια για να καταλαβαίνει ο κόσμος καλύτερα να επιμορφωθεί ως προς τα χρηματοοικονομικά. Και μετά πρέπει να δούμε ότι δεν πρέπει να πληγεί η εμπιστοσύνη στο ευρώ. Αυτό θα γίνει για μένα σαφής προτεραιότητα αν αναλάβω. Θα προσπαθήσω να το ε, προβάλλω όχι μόνο στη Γερμανία και σε άλλες χώρες, το συζητήσαμε και στις κάτω χώρες, το συζητήσαμε σε άλλο επίπεδο, σε άλλες χώρες Εάν σκεφτείτε τι έγινε πριν από ένα-δύο χρόνια με την κρίση του ευρώ, υπήρχε πάλι ένα σοβαρό επίπεδο παρανόηση σε σχέση με το τι κάνει η ΕΚΤ. Δεν θα είμαι λοιπόν Γερμανίδα εκπρόσωπο στην ΕΚΤ, αλλά θα είμαι υπεύθυνη για την Ευρωζώνη συνολικά. Οπότε πιστεύω ότι οι αρμοδιότητε επικοινωνία θα πρέπει να αφορούν ολόκληρη την Ευρωζώνη ταυτόχρονα. Βεβαίω δεν ξέρω αν μπορεί να τα κάνει ένα άνθρωπο αυτά μόνο του, αλλά αυτό που εγώ θα κάνω ω μονάδα είναι να αναζητήσω και ψηφιακού διάβλου. Η ΕΚΤ έχει αυτή τη στιγμή πολύ ωραία επεξηγηματικά σημειώματα στο ιστότοπο ε, είναι πολύ ωραία, αλλά παρά είναι περίπλοκα ακόμα. Ο κόσμος θέλει απλώ να καταλάβει. Συνεχίζουν να απευθύνονται περισσότερο σε οικονομολόγου ε, και γνώστε τη οικονομία παρά στο ευρύ κοινό. Πρέπει λοιπόν ο κόσμο να καταλαβαίνει τι κάνουμε και να ωφελείται. Ευχαριστούμε πολύ. Από τους πράσινους, Λίνας. Ευχαριστώ. Πραγματικά με ξεπλάγει από τον ενθουσιασμό σας, τη δέσμευσή σας. Ε, άκουσα βέβαια και τις απαντήσεις τις ερωτήσεις σας ε, για τις έρευνές σας όσον αφορά τα τελευταία 400 χρόνια κρίσεων στην ιστορία. Ε, μιλάτε πολύ για τις ευπάθειες που έχει το οικονομικό σύστημα. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα ε, πιστεύετε ότι με την τραπεζική εποπτεία έχουν διορθωθεί πράγματα ή με τα, τις διάφορες κλασματικές προσεγγίσεις που έχουμε υιοθετήσει όσον αφορά ε, διάθεση κεφαλαίου, δανείων κτλ. Νομίζετε ότι έχουμε καταφέρει κάτι? Γιατί και οικονομολόγοι άλλοι εξετάζουν την ιστορία και ένας συγκεκριμένο που διάβασα μιλάνε επίσης για ευπάθειες αλλά μιλούν και για, τις, ε, ε, για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που ευθύνονται. Ε, συμφωνείτε? διότι το θέμα της σταθερότητας της οικονομίας εξαρτάται από πολύ περισσότερα πράγματα και έτσι κι ήδη από το 1886 έχουμε αρχίσει να μελετάμε αυτά τα θέματα. Και ο συγκεκριμένο ο οικονομολόγος λέει ότι εξαρτάται τον ισολογισμό από πώ τον κοιτάει κανεί, Οι κυβερνήσεις όταν δανείζονται δεν μπορούν να επιστρέψουν τα δάνεια τα οποία έχουν χρηματοδοτήσει, κάτι το οποίο οδηγεί σε πληθωρισμό. Οπότε, Μπορείτε να σχολιάσετε για τις ευπάθειες αυτές και πιστεύετε ότι μπορεί κάτι να βοηθήσει. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Όλη μου την ακαδημαϊκή ζωή ε, τα μελετάω αυτά. Θα μπορούσα να σας μιλάω για ώρες, αλλά δεν έχω χρόνο, οπότε θα επικεντρωθώ σε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Πρώτον, τι είδους ευπάθειες διαπιστώνουμε. Ε, διαπιστώνουμε όσον αφορά τη σταθερότητα τιμών, κυρίως στην αγορά στέγασης. Βλέπουμε επίσης αλλαγές στη λικτικότητα στον τραπεζικό τομέα και αυτό που εμένα με απασχολεί πιο πολύ είναι ότι αυτό σε ορισμένες χώρες οδηγεί σε ουσιώδεις κινδύνους επιτοκίων. Γιατί εντάξει δεν λέω ότι θα συμβεί, μπορεί όμως να συμβεί κάποια στιγμή. Αυτό θα ήταν πρόβλημα για τις τράπεζες που έχουν δάνεια με ε, πολύ αργότερα ημερομηνία λήξης. Αλλά δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο τις τράπεζες, πρέπει να σκεφτόμαστε και τις ασφαλιστικές εταιρείες που και αυτές αγωνίζονται με τα χαμηλά επιτόκια και που δυσκολεύονται να πληρώσουν τις εγγύσεις που πρέπει να πληρώσουν. Το ίδιο ισχύει και μετά στα εξωδιωτικά ταμεία. Είναι θέμα ρευστότητας τελικά. Βέβαια έχουν περιοριστεί και οι ανταμοιβέ σε αυτούς που αναλαμβάνουν μεγάλα ρίσκα. Και για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια εισήγαμε πάρα πολλές ρυθμίσεις. Ο οικονομικός τομέας σίγουρα είναι πιο ανθεκτικός σήμερα. Έχουμε κάνει πολλά για τον τραμεζικό κλάδο, λιγότερα για τους υπόλοιπους. Πάντως, στη Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή του Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, το βλέπουμε από την τελευταία τους έκθεση, ότι αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ μπερδεμένα και πολύ ακριβά επίσης. Στοιχίζουν. Και γι' αυτό θα πρέπει να τα ξαναδούμε. Εγώ θα προτιμούσα να είχαμε υψηλότερες κεφαλαϊκές απαιτήσει και λιγότερο περίπλοκες ρυθμίσεις. Δεν ξέρω αν οι ίδιες οι τράπεζες θα κάνουν μια τέτοια πρόταση, γιατί αυτό θα τις εξυπηρετούσε σίγουρα. Τώρα για τους οργανισμούς αξιολόγηση πιστοληπτικής εικονότητας. Έχετε δίκιο. Το θέμα της ηθικής εδώ υπάρχει. Τώρα, Μίνσκι. Ο Μίνσκι είναι αυτός ο οποίος έχει επηρεάσει όλη τη λογοτεχνία για τους διάφορους ε, κύκλους. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που έχει γράψει. Θα μπορούσα να είχα μιλήσει περισσότερο για την μακροπροληπτική ε, προσέγγιση, αλλά πάντως είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτά τα οποία έλεγε ο Μίνσκι. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Κούναρ Πέκ από το ID. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα κυρία Σνάμπελ. Δεν ε, είμαι βέβαιος αν κάνατε ε, καλή αρχή. Μέσα του Νοεμβρίου ε, καλέσατε Γερμανούς εμπειρογνώμονες στην οικονομία να διασκεδάσουν τις ε, επικρίσεις τους ε, στις πράξεις ε, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που ήταν και λάθος διότι απειλούν το ευρώ. Ακόμα και ο ΣΑ Ε, θεωρεί ότι, έχει απο... ότι απέτυχε ο Μάριο Ντράγη ε, με τα μέτρα του. Η, Ευρωπαϊκή... η Ευρωζώνη μαζί με την ε, Ιαπωνία έχουν τα χαμηλότερα επίπεδα ανάπτυξης στον κόσμο και το χάσμα πλουσίων και φτωχών είναι μεγαλύτερο από ποτέ. Ε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παραδέχτηκε ότι η πολιτική ποσοτική χαλάρωσης έχει οδηγήσει σε ε, μεγαλύτερα χρέη ε, σε χώρες και επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν κρίση και οι πιο αδύναμες τράπεζες, λέει η έκθεση, συνεχίζουν να είναι πιο ευάλωτες από ό,τι πριν την ποσοτική χαλάρωση. Ε, αυτές οι βλαβερές ε, και ψευδείς ε, ειδήσει που είπατε ότι θα πρέπει να διασκεδαστούν Ε, μήπως προέρχονται από την ίδια Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και κατά τη γνώμη σας πού βρίσκεται το όριο ανάμεσα στις ευλαβερές και ψευδείς ε, ε, ειδήσει και την δικαιολογημένη κριτική. Μπορείτε να μου δώσετε παραδείγματα. Και δεύτερη ερώτηση, μήπως μπορείτε να σχολιάσετε και σύντομα το εξής. Σύμφωνα με μελέτη της τράπεζας DZ, η Γερμανία αποταμιευτές τα τελευταία ε, τα τελευταία χρόνια 648 ε, ε, εκατομμύρια ευρώ έχασαν σε τόκους οι Γερμανοί. Ε, εσείς αναφερθήκατε σε οικονομικά αγράμματους ανθρώπους. Αυτό δεν δείχνει κάποια έπαρση από πλευρά σας. Σας ευχαριστώ κύριε Μπέκε. Θα απαντήσω στα αγγλικά. Ε, ποια είναι τα ψευδή αφηγήματα. Κατά τη γνώμη μου είναι ένα αφήγημα, μια είδηση που αγνοεί ε, τις ε, βασικές οικονομικές γνώσεις ή θεσμικά γεγονότα. Αυτό δεν ε, σημαίνει, και το είχα τουιτάρει και αυτό, ότι δεν θα πρέπει κανείς ε, να ε, επικρίνει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και εγώ το έχω κάνει αυτό η ίδια πολλές φορές και νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό. Νομίζω μάλιστα ότι είναι μέρος της υποχρέωσης λογοδοσίας της. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θα πρέπει όμως να κρίνουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε θέματα που δεν αληθεύουν. Μου ζητήσατε παραδείγματα. Παράδειγμα ψευδούς αφηγήματος είναι ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, ε, απαλωτριώνει τον ε, Γερμανό αποταμιευτή. Αυτό είναι λάθος, διότι η απαλωτρίωση από μόνη της ε, είναι όρος μη θεμητός στο πλαίσιο αυτό και δεύτερον δεν είναι ευθύνη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να δίνει υψηλά επιτόκια στου ε, αποταμιευτέ. Ε, ε, η Υποχρέωση τη είναι να διατηρεί τη σταθερότητα των τιμών. Υπάρχουν πολλά άλλα παραδείγματα. Αυτά που αναφέρατε εσεί είναι οι παρενέργειε τη οικονομική, της νομισματική πολιτική και φυσικά πρέπει να συζητώνται και όπω αναφέρθηκε αυτό συζητιέται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, συζητιέται και στην έκθεση χρηματοοικονομικής σταθερότητα και νομίζω ότι αυτό θα γίνεται όλο και περισσότερο στο μέλλον. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και εγώ η ίδια ανησυχώ όσον αφορά τι παρενέργειε, ιδιαίτερα όσον αφορά την ε, χρηματοοικονομική σταθερότητα. Θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας το θέμα αυτό και δεν έχει καμία σχέση αυτό με αφηγήματα που θα πρέπει να διασκεδαστούν. Ε, αυτά τα αφηγήματα είναι ε, τα ψεύδη που θα πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε ότι είναι ψευδή. Όσον αφορά την έκθεση της τράπεζας DZ, δεν πρόκειται για αναλυθή στοιχεία, πρόκειται για μη πλήρη στοιχεία, διότι αν σκεφτούμε το θεσμικό αντίκτυπο της ε, ε, νομισματικής πολιτικής, ε, δεν θα πρέπει να εξετάσουμε μόνο τους αποταμιευτές, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι και εργαζόμενοι, δηλαδή αν η νομισματική πολιτική έχει σταθεροποιητικό αποτέλεσμα για την αγορά και δεν χάσουν τη, τη δουλειά τους οι άνθρωποι αυτοί, αυτό είναι θετικό αποτέλεσμα για τους ε, πολίτες. Και αν θέλουμε να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα του πώς η νομισματική πολιτική επηρεάζει τους ανθρώπους, θα πρέπει να εξετάσουμε μαζί όλα αυτά τα αποτελέσματα. Θα υπάρχει ετερογένεια, διότι γνωρίζουμε ότι οι ανθρώποι διαφορετικής ηλικίας ε, θα επηρεαστούν σε διαφορετικό βαθμό. Ε, οι οφειλέτες και οι πιστωτές θα επηρεαστούν διαφορετικά, αλλά δεν ε, είναι αλήθεια ότι ε, υποφέρουν περισσότεροι στοχότεροι, διότι ε, αυτοί δεν έχουν πολλές αποταμιεύσεις. Είναι όμως πιθανότατα οι άνθρωποι που βρήκαν δουλειά επειδή η οικονομική ανάπτυξη ήταν πιο μεγάλη από ότι, από με άλλη νομισματική πολιτική. Ευχαριστώ το ECR. Ο κύριος Φαν Όβερτφελτ. Ευχαριστώ κυρία Σνάμπελ, ευχαριστώ που είστε εδώ. Προηγουμένως κάνατε μια δήλωση και είπατε ότι είναι πολύ λίγοι αυτοί που πραγματικά καταλαβαίνουν τι συμβαίνει. Το βρίσκω αξιοσημείωτο και πραγματικά με όλο το σεβασμό διαφωνώ. Νομίζω ότι ήρθε η στιγμή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι κάποιες φορές το να χρησιμοποιεί πολύ ε, μυστικιστική και απόκριφη γλώσσα ε, συμβάλλει στο να μην γίνεται και κατανοητή τις επικοινωνιακές σας δεξιότητες ελπίζω να τις βελτιώσετε εσείς οι ίδια. Και έχω δύο ερωτήσεις επιπλέον. Ε, κυρία Λαγκάρντο, ο κύριος Πανέτα και εσείς οι ίδια αναφερθήκατε συχνά στις παρενέργειες της νομισματικής πολιτικής. Θα ήθελα να μου πείτε ποιες είναι οι βασικές δύο παρενέργειες που σας ανησυχούν περισσότερο σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη χρονική στιγμή. Και η δεύτερη ερώτησή μου έχει να κάνει με τις κλιματικές αλλαγές, την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Η κυρία Λαγκάρτα το όρισε ως μια προτεραιότητα κρίσιμη για την αποστολή που αναλαμβάνει. Ο κύριο Γέιτμαν τη Bundesbank, τη Ομοσπονδιακή Τράπεζα τη Γερμανία, ταυτόχρονα είπε το εξή και πάλι δήλωση που θα διαβάσω, νομισματική πολιτική η οποία επιδιώκει συγκεκριμένα περιβαλλοντικού στόχου, μπορεί να ε, είναι υπερφορτωμένη με πολλού στόχου. Ήθελα λοιπόν και τη δική σα τοποθέτηση επί του θέματο. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις αυτές. Πολύ σύντομα για την πρώτη παρατήρηση νομίζω ότι έχετε το δίκιο. Η επικοινωνία της νομισματικής πολιτικής στο παρελθόν ήταν πολύ τεχνική ε, και γραφειοκρατική. Πρέπει να μιλάμε όχι πλέον στους γνώστες, στις αγορές, αλλά και στο ευρύ κοινό. Και πρέπει να γίνει αυτό με έναν τρόπο ε, ε, μη γραφειοκρατικό. Υπήρξα δασκάλα για πολλά χρόνια και ξέρω πώς πρέπει να γίνει αυτό. Υπάρχει ένα επίπεδο εκλαίκευσης, απλούστευσης, που δεν θα είναι πάντα όλα 100% σωστά, αλλά πρέπει να πάψουμε να κινούμαστε μόνο σε ένα τεχνικό επίπεδο αυστηρά. Πρέπει να τα απλοποιήσουμε. Και για τη δεύτερη παρατήρηση, δύο σημαντικότερες παρενέργειες. Θα έλεγα η πρώτη είναι η οικονομική σταθερότητα και η δεύτερη, ο αντίκτυπος στους αποταμιευτές. Ε, οι οικονομίες τους είναι το θέμα. Γιατί πολιτικός αυτό θα είναι μείζον θέμα. Ε, δεν είναι ακριβώ μέρο τη εντολή του ΕΚΤ να προσφέρει εγγύηση για του αποταμιευτέ, όμω είναι μείζον πολιτικό θέμα και θα πρέπει να το φροντίσουμε. Πρέπει βεβαίω να έχουμε υπόψη και το γεγονό ότι όταν μιλάμε για χαμηλά επιτόκια, αυτό δεν αφορά μόνο την ΕΚΤ, όπω είπα και στην εισαγωγική μου ομιλία. Αυτό οφείλεται και σε άλλες τάσεις ε, χαμηλής ανάπτυξης και κυρίως αυτά της παραγωγικότητας. Στην παραγωγικότητα η ΕΚΤ δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Πρέπει οι κυβερνήσεις να χαράξουν πολιτικές στραμμένες προς το μέλλον, να στηρίξουν την εξέλιξη και την καινοτομία προκειμένου να τονωθεί η παραγωγικότητα και με αυτόν τον τρόπο να αυξηθούν τα επιτόκια η ΕΚΤ με την νομισματική της πολιτική αυτό μπορεί να το υποστηρίξει. Αλλά όπως είπα στην αρχική μου δήλωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις διευθυντικές πολιτικές των κυβερνήσεων. Αυτό είναι ζωτική σημασία, αυτό το θυμόμαστε. Παρ' όλα αυτά παραμένει σημαντικό. Για τις κλιματικές αλλαγές Κοιτάξτε, οι κλιματικές αλλαγές είναι το ένα και σημαντικότερο ζήτημα που μας απασχολεί σήμερα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Επίσης, τελείως σαφές είναι ότι ο καθένας πολιτικός ευθύνων πρέπει να σκεφτεί τι μπορεί να κάνει σε σχέση με τις κλιματικές αλλαγές. Η Κεντρική Τράπεζα δεσμεύεται από την εντολή τη Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει τα πάντα και βεβαίω οι κλιματικέ αλλαγέ δεν είναι μέρο τη πρωταρχική εντολή τη. Έκτη είναι σταθερότητα των τιμών. Βεβαίω, δεύτερο γενός μπορεί να υποστηρίξει την οικονομική πολιτική συνολικά η ΕΚΤ. Οι κλιματικέ αλλαγέ λοιπόν μπορεί να είναι μέρο των στόχων τη οικονομική πολιτική. Αλλά μόνον εφόσον δεν έρχεται σε αντιδιαστολή με τον πρωταρχικό στόχο τη εντολή. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Η νομισματική πολιτική μπορεί να ε, κάνει κάτι, αλλά όχι τα πάντα. Είναι περιορισμένη. Πρέπει κανείς να τονίσει ότι η ΕΚΤ δεν θα είναι το θεσμικό όργανο που θα ασχολείται πραγματικά με τις κλιματικές αλλαγές. Αυτό πρέπει να το κάνουν οι κυβερνήσεις. Χρειάζεται ένα συνολικό σύστημα τιμολόγησης του άνθρακα, των δικαιωμάτων ε, εκπομπών δηλαδή. Αυτό όμως δεν μπορεί να το αποφασίσει η ΕΚΤ. Ε, μπορεί να κάνει πολλά, αλλά όχι αυτό. Αλλά αυτά ως προς την απάντησή μου. Ευχαριστούμε ο κύριος Σίρντεβαν από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Σνάμπελ. Μας είπατε κάποια στοιχεία και για το πολιτικό σας πρόγραμμα. Το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον και την όλη συζήτηση. Θα ήθελα και εγώ να συνεισφέρω ε, λοιπόν με τις δικές μου παρατηρήσεις. Η κυρία ε, Λαγκάρτ, χθε στον πολιτικό μας διάλογο στην ΕΚΟΝ, είπε ότι πρέπει να υπάρξει μια αναθεώρηση της πολιτικής στρατηγικής ε, για τα νομισματικά θέματα στην ΕΚΤ. Εσείς βλέπετε ότι αυτό είναι απαραίτητο Και πώς θα γίνει αυτή η αλλαγή στο στατικικό προσανατολισμό της ΕΚΤ στο επίπεδο το νομισματικό. Και η δεύτερη ερώτηση που τονίσατε, η σταθερότητα των τιμών είναι το πρωτογενέ, η πρωτογενής εντολή της ΕΚΤ. Όμως ε, και η οικονομική ανάπτυξη και η τόνωση της βιωσιμότητας του οικονομικού συστήματος είναι ένα θέμα και με άλλους πολιτικούς στίχους, ε, στόχους που καλλιεργούνται και, από και επιδιώκονται από άλλες κεντρικές τράπεζες. Όπως ένας εξισορροπημένος ισολογισμός. Ε, η ΕΚΤ θα το λάβει αυτό υπόψη στην αναθεώρηση της στρατηγικής πολιτικής για τα νομισματικά. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. στην νομισματική πολιτική, στην αναθεώρηση τη ε, νομισματική στατική πολιτική. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε με στην εντολή μα. Δεν είναι δουλειά μα να αλλάζουμε εντολή. Πρέπει να πάρουμε την εντολή όπω μα έχει δοθεί. Νομίζουμε λοιπόν ότι βάσει αυτή τη εντολή κάνουμε καλή δουλειά. Δεν θα ξεκινήσω τώρα μια συζήτηση περί αλλαγή τη εντολή μα. Δική σα ευθύνη είναι, όχι τη ΕΚΤ. Νομίζω η αναθεώρηση τη στρατηγική πολιτική για τα νομισματικά είναι πολύ σημαντική. Η ΕΚΤ έχει κάνει μόνο μία πολιτική αναθεώρηση και αυτό έγινε πριν από πάρα πολύ καιρό, το 2003. Έκτοτε έχουν γίνει πολλά και η οικονομία έχει αλλάξει εκβάθρων. Και η νομισματική πολιτική έχει αλλάξει επίσης. Νέα εργαλεία αναδύθηκαν ο κόσμος που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι πολύ διαφορετικός από τότε. Τότε όλοι ανησυχούσαν για τον υπερβολικό πληθωρισμό. Θα θυμάστε την τότε συζήτηση. Η ε, έπρεπε να ακολουθήσει το μοντέλο της Bundesbank, διότι νόμιζαν τότε ότι η Bundesbank αγκιάται τον χαμηλό πληθωρισμό. Τώρα έχουμε την ανάποδη απειλή. ο πολύ χαμηλός πληθωρισμός Και έπρεπε να δούμε ότι οι μηχανισμοί στους οποίους επαφιόμαστε ως τώρα λειτουργούν διαφορετικά. Πρέπει να σκεφτούμε και την καμπύλη Φιλίπς, ε, την σχέση απασχόλησης πληθωρισμού ας πούμε. Υπάρχουν λοιπόν εντατικέ συζητήσει σε επιστημονικό, σε, ε, ε, σε πανεπιστημιακό επίπεδο για το τι γίνεται με αυτή την καμπύλη, αν έχει διακοπεί και στρεβλωθεί, αν ε, απλώ αμβλύνεται. Τέλο πάντων, όλα αυτά πρέπει να τα καταλάβουμε καλά, να τα μελετήσουμε. Πρέπει να γίνει μια διεξοδική αναθεώρηση βάσει των επιστημονικών στοιχείων των πανεπιστημιακών πορισμάτων θα μπορούσαν εκείνοι να αναλάβουν ένα μέρος της δουλειάς που πρέπει να προηγηθεί για να δούμε πώς ακριβώς λειτουργούν τα εργαλεία μας, ποιες είναι οι παρενέργειες, Ε, ήταν ένα σημαντικό στοιχείο της πολιτικής αναθεώρησης Ποια είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τα επιτόκια, τι σημαίνει αυτό για τους στόχους του πληθωρισμού και μόνο μετά από μια τόση, τόσο προσεκτική και διεξοδική ανάλυση μπορούμε να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Μπορεί στο τέλος να μην χρειαστούν τόσο μεγάλες προσαρμογές. Δεν είναι ξεκάθαρο ότι θα πρέπει στο τέλο να τα φέρουμε τα πάνω κάτω στο όλο σύστημα. Δεν νομίζω να χρειάζεται αυτό. Ε, θα χρειαστούν ίσως κάποιες διευκρινήσεις, κάποιες μικροπροσαρμογές. Κατά πάσα πιθανότητα το βασικότερο θέμα θα είναι πώς να ενσωματώσουμε άλλους στόχους και οι σημαντικότεροι θα είναι οι κλιματικές αλλαγές. Πώς λοιπόν να το κάνουμε χωρίς να ξεφύγουμε από την εντολή μας και χωρίς να θέσουμε να αμφιβόλο την ανεξαρτησία μας. Αυτό θα πρέπει να μας οδηγήσει γενικώ στην αναθεώρηση της ε, πολιτικής μας. Δεν θα πρέπει να υπάρξει καμία αμφιβολία για την ανεξαρτησία της ΕΚΤ στην εντολή τη. Ευχαριστούμε κυρία Χούμπνερ από το ΕΛΚ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Μία ερώτηση έχω πρώτα απ' όλα για το διεθνή ρόλο της Ευρώπης. Θα συμφωνήσετε μαζί μου φαντάζομαι ότι ποτέ στην ιστορία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, από την αρχή του ευρώ δηλαδή, δεν υπήρχε πρόθεση ενίσχυσης του διεθνούς ρόλου ε, της Ευρώπης. Υπήρχαν διάφοροι λόγοι και σίγουρα ένας από αυτούς ήταν η ανησυχία ότι η χρήση του νομίσματος διεθνώς θα δημιουργούσε πιέσει στην νομισματική πολιτική της ΕΚΤ, γιατί η κατάσταση θα ήταν διαφορετική. Τώρα όμως βλέπουμε ότι αλλάζουν τα πράγματα. Το ακούσαμε και από την ε, Επιτροπή ότι αλλάζει η κατάσταση. Τι νομίζετε λοιπόν ε, για αυτό το θέμα, το να έχουμε δηλαδή ένα περισσότερο ισχυρό διεθνώς ευρώ και ποιος ο ρόλος της ΕΚΤ σε αυτή την περίπτωση, εφόσον όντως ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο. Η δεύτερη ερώτησή μου έχει να κάνει με την ε, Εκτελεστική Επιτροπή. Ε, ε, θα ήθελα να μου πείτε, μετά από την ερώτηση και του κύριου Φέμπερ, που εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο προχωρούν τα πράγματα, συγγνώμη, στο Διοικητικό Συμβούλιο, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Από ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχει αρκετή διαφάνεια στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εξαρτάται βέβαια από το με ποιον συναντιόμαστε, αλλά αυτή είναι η εμπειρία μας πάντως. Και ακούμε από καιρού καιρό ότι γίνονται προσπάθειες στο Διοικητικό Συμβούλιο από πλευρά των μελών του δηλαδή να πιέσουν την ΕΚΤ για την νομισματική της πολιτική. Οπότε ρωτάω αυτή τη σχέση πώς την εκτιμάτε εσείς. Πιστεύετε κι εσείς ότι θα έπρεπε να αλλάξουν οι διαδικασίες που χρησιμοποιεί η ΕΚΤ και θα ήσασταν έτοιμοι να μας δίνετε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ΕΚΤ. Έπειτα, πιστεύετε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν θα έπρεπε να είναι λίγο περισσότερο διαφανές απέναντί μας και τέλος πάντων τι όρια βάζετε εσείς αυτή τη διαφάνεια. Ευχαριστώ. Απάντηση. Σας ε, ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως. Αυτό είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Ο διεθνής ρόλος του ευρώ δηλαδή. Και συμφωνώ μαζί σας ότι πριν από μερικά χρόνια δεν είχαμε και πολύ όρεξη να συζητάμε γι' αυτό. Αλλά η αλλαγή οφείλεται και ε, στην γεωπολιτική κατάσταση που έχει επίσης αλλάξει ριζικά. Οπότε στην Ευρώπη αντιλαμβανόμαστε διαφορετικά τα πράγματα και πιστεύουμε πια ότι η Ευρώπη πρέπει να παίξει έναν περισσότερο ισχυρό ρόλο στην Ευρώπη. Και το νόμισμα εννοείται ότι αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, δεν είμαι και τόσο σίγουρη <clears throat> για το πόσο πολύ θα ήθελα ε, να τονίσω αυτό το στόχο Πάντως σίγουρα έχει να κάνει και με την γενικότερη συζήτηση για τα ασφαλή περιουσιακά στοιχεία, που γίνεται και σε άλλα πλαίσια. Ένα πλαίσιο είναι μεταρρύθμιση στην Ευρωζώνη. Έχουμε τη συζήτηση για το έντις, για την ε, έκθεση ε, σε δημόσιο χρέος ότι υπάρχει αποσταθεροποίηση στη συνέχεια και κάποιοι λένε ότι το ευρωπαϊκό ε, ακριβώς ασφαλές ε, αυτό περιουσιακό στοιχείο ε, αποτελεί και αυτό στο οποίο μπορούμε να βασιστούμε για τα πάντα. Πάντως πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ καλά το θέμα της αμοιβοποίησης του επιμερισμού του κινδύνου. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε μια ένωση κυρίαρχων κρατών. Αν λοιπόν υπάρξει ασφαλές ε, περιουσιακό στοιχείο, όπως το ονομάζουμε, θα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει επιμερισμός κινδύνου. Οπότε δεν βλέπω πώς ακριβώς θα μπορούσε να γίνει. Τέλος, για το Διοικητικό Συμβούλιο. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι υπάρχει ήδη πολύ μεγάλη διαφάνεια στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δείτε τους λογαριασμούς, εγώ πιστεύω ότι είναι με μεγάλες λεπτομέρειες. Αυτό που δεν έχετε και ίσως αυτό είναι που ζητάτε, είναι ότι δεν ξέρετε ποιος ψήφισε τι. Πόσοι ψήφισαν, ποιοι ήταν υπέρ, ποιοι... Εγώ εδώ είμαι βέβαια προβληματισμένη, γιατί το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι οι επικεφαλείς των κεντρικών τραπεζών θεωρούνται μερικές φορές σαν να εκπροσωπούν τις χώρες τους. Κάτι το οποίο όμως είναι καταστροφικό. Δεν πρέπει να είναι έτσι όλοι εκπροσωπούν την Ευρωζώνη συνολικά. Αν λοιπόν υπάρχει ψηφοφορία και η ψηφοφορία αυτή αποκαλυφθεί στο κοινό, πιστεύω ότι η πολιτική πίεση τότε στα επιμέρους μέλη θα είναι μεγάλη και δεν νομίζω ότι είναι μια καλή ιδέα να γίνει κάτι τέτοιο. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μπέλκα από τους Σοσιαλδημοκράτες, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις έχω. Ο Μάριο Ντράγκη είπε ότι αναφέρθηκε στις θέσεις απασχόλησης και το ε, εισόδημα των εργαζομένων και δεν είμαι καν βέβαιος αν ε, το είπε αυτό, αλλά ε, αυτή η αντίθεση γίνεται από πολλούς παρατηρητές. Εσείς πώς βλέπετε την αντίθεση αυτή, ότι ή το ένα θα έχουμε ή το άλλο. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αγωνίζεται όσο πιο καλά μπορεί να επαναφέρει τον πληθωρισμό κοντά στο 2%. Όπως ε, και η Τράπεζα της Ιαπωνίας. Πόσο διαφέρει από τη Ιαπωνία η Ευρωζώνη. Γιατί πιστεύουμε ότι εμείς μπορούμε να πετύχουμε την αύξηση του πληθωρισμού. Σας ευχαριστώ. Ωραία. Λοιπόν, όσον αφορά την πρώτη σας παρατήρηση, ήδη αναφέρθηκα εν μέρη σε αυτό. Από τη σκοπιά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, δεν πρόκειται για αντίθεση, δεν πρόκειται για ε, κάτι που πρέπει να διαλέξουμε ένα από τα δύο, διότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, έχει ως καθήκον την ε, διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, πράγμα που επηρεάζει ένα σωρό άλλους τομείς και η νομισματική πολιτική ε, πάντα έχει συνέπειες. Όσον αφορά την ανακατανομή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όμως δεν έχει εντολή για ανακατανομή. Δεν μπορεί να αποφασίζει ποιος κερδίζει και ποιος χάνει. Και γι' αυτό οι συνέπειε όσον αφορά την κατανομή είναι φυσική συνέπεια της νομισματικής πολιτικής. Οι συνέπειε όμως θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε πολιτικό επίπεδο. Για παράδειγμα, εάν σκεφτούμε τα χαμηλά επιτόκια και αναφέρομαι στη συζήτηση που γίνεται εντός της Γερμανίας, Γνωρίζουμε ότι ταυτόχρονα έχουν εξοικονομήσει πολλά χρήματα οι κυβερνήσεις. Οι κυβερνήσεις λοιπόν είχαν κέρδος επειδή ε, ε, έχουν υψηλό χρέος, ε, πλήρωναν λοιπόν πολύ χαμηλότερους τόπους, τόκους και η Κεντρική Τράπεζα στο, τελικά δεν επιτρέπεται να λαμβάνει την απόφαση ποιος θα χάνει και ποιος θα κερδίζει από την οικονομική κατάσταση. Δεν είναι κάτι που εμπίπτει στην εντολή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όσον αφορά την σύγκριση ανάμεσα στη ζώνη του ευρώ και τη Ιαπωνία, σίγουρα υπάρχουν κάποιες ομοιότητες, μία εκ των οποίων ε, είναι ότι υπήρξε μια βαθιά τραπεζική κρίση στην αρχή του προβλήματος. Επίσης ε, υπάρχουν κάποια διαρθρωτικά στοιχεία όπως είναι η δημογραφική αλλαγή. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα και στη Ιαπωνία και στη ζώνη του ευρώ. Πέρα από αυτά όμως ε, η θέση της Ιαπωνίας και η θέση της Ευρωζώνης ε, διαφέρουν διότι η Ιαπωνία είναι κυρίαρχο κράτος με δική της κεντρική τράπεζα ενώ η Ευρωζώνη είναι μια νομισματική ένωση. Αυτό έχει πολλές συνέπειες. Σημαίνει ότι πρέπει να είναι κανείς ιδιαίτερα προσεκτικός κατά τη σύγκριση ε, των δύο αυτών ε, καταστάσεων. Η Ευρωζώνη έχει εφαρμόσει πολλές μεταρρυθμίσεις για να αντιμετωπίσει την ε, αβεβαιότητα που διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης. Η Τραπεζική Ένωση είναι πολύ σημαντικό στοιχείο και σε παγκόσμιο επίπεδο είδαμε μια πολύ ε, αποφασιστική αντίδραση. Ε, είδαμε ότι ε, ελήφθησαν μέτρα για ενίσχυση του τραπεζικού τομέα, κάτι που στη Ιαπωνία καθυστέρησε πολύ περισσότερο. Επίσης υπάρχει το πρόβλημα του προβλήματος του δημοσίου χρέους ε, στην Ευρωζώνη, κάτι που δεν ε, αντιμετωπίζει η Ιαπωνία. Η Ιαπωνία έχει υψηλό δημόσιο χρέος, ε, αλλά βιώσιμο από ό,τι φαίνεται. Είναι λοιπόν πολύ διαφορετικές οι καταστάσεις και εγώ δεν θα τις συνέκρινα άμεσα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε τις ερωταπαντήσεις και ευχαριστώ τους συναδέρφους μου και ευχαριστώ και σας κυρία Σνάμπελ. για την ακρόαση αυτή. Μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης σε λίγα λεπτά για να ε, επιτρέψουμε αλλαγή σκηνικού. Okay. I would move to the next... Λοιπόν, περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη, που είναι η παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης 2019 για την Τραπεζική Ένωση. Είναι η ετήσια έκθεση μετά την τέταρτη η οποία κάλυψε το 2018 τις εξελίξεις στη Τραπεζική Ένωση και εγκρίθηκε και από την Ολομέλεια. Στόχος της έκθεσης αυτής είναι να δούμε ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στην Τραπεζική Ένωση από τότε που ανέλαβε το ρόλο του ενιαίου επόπτη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αφού ανέλαβε τα πλήρη καθήκοντά του τον Ιανουάριο 2016 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου. Ήδη εξετάστηκαν οι πρώτες περιπτώσεις το καλοκαίρι του 2017. Η έκθεση αυτή πρέπει να εξεταστεί επίσης και υπό το φως νομοθετικών προτάσεων για ε, την τελειοποίηση των κανόνων της Βασιλείας 3 και μετά και από την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπής για το ΕΔΙΣ, δηλαδή το Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων και εν ώψη της ολοκλήρωσης ε, της Τραπεζικής Ένωσης. Ο εισηγητής είχε 7 συναντήσεις με τις αρχές και τους ενδιαφερόμενους, όπου είχαν προσκληθεί όλες οι ομάδες και όλες και όλες οι εισηγητές. Όπως κάναμε και τα προηγούμενα χρόνια και εδώ καλύπτουμε πολλά και διάφορα θέματα σε τέσσερα κεφάλαια, η γενική εποπτεία, η ασφάλιση κλπ. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο τώρα στον εισηγητή τον ε, Πέδρο Μάρκες από τους Σοσιαλδημοκράτες. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι οι πρώτες μου εισαγωγικέ παρατηρήσεις στα πορτογαλικά παρακαλώ και μετά τις ερωτήσεις σας, εντάξει θα τις απαντήσω στα αγγλικά. Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω την Επιτροπή ΕΚΟΝ και τους συνεργάτες της για την υποστήριξη είχαμε τη δυνατότητα να ακούσουμε μια σειρά από ενδιαφερομένους και θεωρώ ότι ήταν σημαντικό αυτό και για τη δική μας τη δουλειά και για τους σκιώδεις στην προετοιμασία αυτής της συζήτησης που έχουμε ξεκινήσει και που τώρα θα κάνουμε. Εδώ κοιτάζουμε τη σημασία του τραπεζικού τομέα για τον οικονομικό κλάδο γενικώ και το βάρος του τραπεζικού τομέα στην Ευρώπη σε σχέση με άλλες περιοχές του κόσμου. Ιδίω της ΕΠΑ. Πράγματι, το τραπεζικό σύστημα, συγκεκριμένα η Τραπεζική Ένωση, μπορεί να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης αρκεί να υπάρξει κατάλληλη υποστήριξη στις επενδύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ταυτόχρονα η αστάθεια του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος μπορεί να ε, εξαρτηθεί από την έλλειψη εμπιστοσύνης ή την έλλειψη επενδύσεων μακροπρόθεσμα. Γι' αυτό ελήφθη η απόφαση να συμβάλλουμε στη δημιουργία της Τραπεζικής Ένωσης και η έκθεση αυτή επισημαίνει τις ε, καλές εξελίξεις ε, του κλάδου αυτού προς την Τραπεζική Ένωση τονίζει πώς πρέπει να υποστηριχθούν οι στόχοι αυτοί ε, μέσα από τα χρόνια, ενισχύοντας την αντοχή του κλάδου. Το 2019 δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιηθούν από κάποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ε, οι διατάξεις του μηχανισμού εξυγένσης. Τα τελευταία χρόνια επίσης τονίζεται πώς πήγε η κερδοφορία των τραπεζικών ε, ιδρυμάτων που βάσει της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής έφτασε σε ικανοποιητικά επίπεδα ο χαμηλός, ε, το χαμηλό επίπεδο κινδύνου και τα χαμηλά επιτόκια έχουν βεβαίως ε, επηρεάσει τον τραπεζικό τομέα στην Ευρώπη. Η έκθεση απαριθμεί και προσπαθεί να κοιτάξει την καλή εξέλιξη των δύο πυλών που έχουν να κάνουν με την υποστήριξη και την, ε, διπλή, την εποπτεία μάλλον και τη διπλή ε, ανακεφαλοποίηση του τραπεζικού τομέα στην Ευρώπη. Ε, στην εποπτεία γνωρίζουμε κάποια από τα πορίσματα, το είπα και σε σχέση με την αθεκτικότητα του τομέα, αλλά και την πολύ γρήγορη εξέλιξη του Ευρωπαϊκού Συστήματο Εξυγίανση Ανακεφαλοποίηση, κάτι που συζητήθηκε ήδη και προετοιμάζει τον τραπεζικό κλάδο για ενδεχομένε μελλοντικέ καταστάσεις ε, προβληματικές, ώστε να είναι πιο εύρωστος. Η έκθεση στη συνέχεια εντοπίζει μια σειρά από προκλήσει για την Τραπεζική Ένωση στο μέλλον, ιδίω για την ολοκλήρωσή τη, κάτι που αναφέρθηκε προηγουμένω και από την Πρόεδρο, αλλά θα πρέπει να το λάβουν υπόψη και άλλοι από του συμμετέχοντε, εκπρόσωποι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή και τη Κεντρική Τράπεζα, που ήδη το έχουν πει. Το να ενισχυθεί η ΕΚΤ είναι μια πρόκληση που να αντιμετωπίσουμε, αλλά και να ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση είναι σημαντικό ώστε οι πυλώνες αυτές να προχωρήσουν με το σύστημα έντις, το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων μεταξύ άλλων. Και θα πρέπει να συμπληρωθεί και από το backstop, το μηχανισμό διασφάλισης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασφαλείων. Εδώ λοιπόν ο τρίτος πυλώνας της Τραπεζικής Ένωσης που έχει σχέση με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό ε, Ασφάλισης των Καταθέσεων, ΕΣΑΚ, θα πρέπει να προχωρήσει και σε ένα σημαντικό στοιχείο ευρωπαϊκής πολιτικής την διασύνδεση μεταξύ των κρατικών συστημάτων και το, ε, των εθνικών, ε, των, ε, του ευρωπαϊκού επίπεδου σε, στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αυτό το είπε και η συνάδελφος Χούμπνερ μόλις προηγουμένως στην ακρόαση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και το European Safe Asset, τα ασφαλή περιουσιακά στοιχεία ώστε να πάυσει αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνη μεταξύ κρατικών συστημάτων και του χρηματοοικονομικού. Επίση, εντοπίσαμε και άλλε προκλήσει και δυσκολίε στην ολοκλήρωση τη Τραπεζική Ένωση, όπω η ανάγκη, ο κατακαιρματισμό που υπάρχει ακόμα στο χρηματοοικονομικό τοπίο τη Ευρώπη, ιδίω στου μηχανισμού ρευστοποίηση στις τράπεζες, SRM και αυτό που αναφέρθηκε και προηγουμένως, το πώς επηρεάζουν οι εταιρείε FinTech το τραπεζικό σύστημα στην Ευρώπη, θα πρέπει να διέπονται από ίδιους κανόνες, όπως και το τραπεζικό σύστημα ε, για τις τραπεζικές υπηρεσίε. Επίσης γίνεται αναφορά στην σημασία της ε, παραοικονομίας στο τραπεζικό κλάδο, ε, το shadow banking θα πρέπει και εδώ αυτό να ληφθεί υπόψη ως φαινόμενο με ένα πλαίσιο ρύθμισης και εποπτείας και για αυτόν τον κλάδο διότι είναι ένα μέσο χρηματοδότησης της οικονομίας αλλά δημιουργεί και ρίσκα, ελοχεύουν κίνδυνοι για, για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας μετά το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και σχετικές πρακτικές είναι στοιχεία που θα πρέπει να τα μελετήσουμε, καθώς και το χρηματοδότηση της τρομοκρατίας για να δούμε την τωρινή κατάσταση. Ε, κίνδυνοι αυτοί δεν έχουν απαλληφθεί και θα χρειαστεί περισσότερη διαφάνεια και περισσότερη ενημέρωση των ε, καταναλωτών για, του, για τους κινδύνους, ε, για την αστάθεια, για το πώς θα πρέπει να εξελιχθεί η ευρωπαϊκή οικονομία. Και αυτό ε, αναφέρεται στην έκθεση για να δούμε κατά πόσον μπορεί να συνεχιστεί η συζήτηση για ένα ευρωπαϊκό οίκο αξιολόγηση στην Ευρώπη και να δούμε κατά πόσο οι δείκτες βιωσιμότητας της χρηματοδότησης μπορούν να ληφθούν απόψη από ένα τέτοιο ευρωπαϊκό οίκο. Στο παρελθόν υπήρχε ευρία συνένεση για τη δημιουργία μηχανισμών ε, πιο κατάλληλων για την αντιμετώπιση των κινδύνων στο ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό σύστημα Χρειαζόταν περισσότερη ανεξαρτησία σε σχέση με αυτή την αξιολόγηση, θεωρούσαμε τότε. Τώρα πρέπει να συνεχίσουμε να κοιτάζουμε διαρκώ κατά πόσον όλε οι προσπάθειε για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κυρίω ο διαχωρισμό των εμπορικών δραστηριοτήτων από αυτέ των επενδυτικών, των επενδύσεων μάλλον, ε, συνάδουν με την ανάγκη να προχωρήσει αυτή η κατάλληλη αξιολόγηση. Πρόεδρε, Λίγο πολύ αυτό είναι το πλαίσιο εντό του οποίου κινείται η έκθεση που έχω αποβάλει. Τώρα βεβαίω θα την κρίνουν οι συνάδελφοι και πρέπει να πούμε ότι η στιγμή για να ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση έφτασε. Ξεκίνησε και η νέα θητεία, τα νέα θεσμικά όργανα, όλοι οι θεσμοί ασχολούνται σοβαρά με τι υποχρεώσει του. Θα πρέπει να προχωρήσουμε στο επίπεδο τη Οικονομική και Νομισματική και νομίζω ότι αυτή ήταν η θέση του Κοινοβουλίου και στο παρελθόν μου φαίνεται απαραίτητο να μην προχωρήσουμε σε μια σταθερή νομισματική πολιτική, πράγμα που δεν είναι και εφικτό, χωρί τραπεζική ένωση. Γι' αυτό λοιπόν η έκθεση αυτή εφόσον εγκριθεί πολιτικώ, θα μα επιτρέψει, επιτρέψει σε όλα τα θεσμικά όργανα να κάνουν σωστά τη δουλειά του. Ευχαριστώ πολύ όλου του συναδέλφου για τι συνεισφορέ του. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Δίνω τώρα το λόγο στους σκιώδεις συγητές που θα έχουν τέσσερα λεπτά ο καθένας. Θα ξεκινήσουμε από την κυρία Χίμπνερ από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή η δουλειά που έχει γίνει και νομίζω ότι ε, τα περισσότερα θέματα που μας ενδιαφέρουν ε, έχουν συμπεριληφθεί. Όπως γνωρίζετε ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά εδώ και χρόνια και υπάρχουν ε, ε, θέματα που ανακύπτουν και θα πρέπει να ανακύπτουν ε, συνεχώς ε, εφόσον δεν έχει, ενοποιηθεί, δεν έχει ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση. Με το ψήφισμά μας θα πρέπει λοιπόν να αναφέρουμε τα μη ξυπηρετούμενα δάνεια, το να γίνει λειτουργική η Τραπεζική Ένωση. Όλα αυτά είναι θέματα που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται. Επίσης ε, θα ήθελα κάποιες ε, προσθήκες στο τελικό κείμενο, την ε, ανάγκη αναθεώρησης του συστήματος κρατικών ενισχύσεων και όσον αφορά τον ανταγωνισμό, αλλά και όσον αφορά το θέμα της αναλογικότητας των μικρών τραπεζών και την καλύτερη σχέση εξυγίανσης ε, και αφαιρεγκαιότητας. Επίσης, ε, όσον αφορά το κατά πόσο είναι και οι ευρωπαϊκές τράπεζες, διότι πρέπει να το δούμε αυτό και ε, σε σχέση με άλλες δικαιοδοσίες. Έτσι μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα δεν είναι ακόμα αυτή που θα έπρεπε να είναι Επίσης, πιστεύω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στην Ένωση Κεφαλαιογορών, καθώς και το ΙΜΙΡΙ και το CCP, διότι βλέπουμε κάποιες ε, αλλαγές στους τομείς αυτούς. Και επίσης, όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού Βασιλεία 2, ε, θα αποτελέσει σημαντικό βήμα στην ολοκλήρωση της ε, τραπεζικής μεταρρύθμισης. Πρέπει όμως επίσης να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη και το θέμα των ε, κεφαλαιακών απαιτήσεων είναι επίσης ένα δύσκολο θέμα. Ε, οι νέοι κίνδυνοι αναφέρονται όπως το κλίμα, υπάρχουν όμως και άλλοι νέοι κίνδυνοι μεγάλης σημασίας. Θα πρέπει να εξετάσουμε επίσης όχι μόνο το κόστος αλλά και τις ευκαιρίες. Και Επίσης, ε, νομίζω ότι θα πρέπει να ε, δούμε και τι παραπάνω μπορεί να γίνει για να ε, ενισχύσουμε τη θέση των ευρωπαϊκών τραπεζών. Ολοκλήρωσα σε λιγότερο από τέσσερα λεπτά. Χαρίζω ένα λεπτό σε κάποιον άλλο μιλητή. Ο κύριος Κέλεχερ από το Ρήνιου. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να επικροτήσω την έκθεση αυτή και να ευχαριστήσω τον Πέτρο Μαρκέση για τις παρατηρήσεις του. Μας ε, ενδιαφέρει η εμπιστοσύνη στην Τραπεζική Ένωση. Είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ε, η ακαιρεότητα και η εμπιστοσύνη στο ευρώ. Η αμοιβαιοποίηση του κινδύνου είναι τομέα κλειδί και θα πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτό. Αυτό φυσικά θα οδηγήσει σε δυσκολίες όσον αφορά την πολιτική της Ευρώπης αυτής καθ' αυτής στο πλαίσιο αυτό τα ε, ασφαλή ε, περιουσιακά στοιχεία, τα safe assets είναι ένα θέμα με το οποίο θα πρέπει να ασχοληθούμε άλλα. Ε, στο Ίκρη e θα υπάρχουν πολιτικές δυσκολίες ε, στο Συμβούλιο και αλλού. Νομίζω όμως ότι πρέπει να συνεχίσουμε να ακολουθούμε τον δρόμο αυτό, διότι ε, αν ε, θέλουμε να... Εάν είμαστε σοβαροί όταν μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Αγγίσης, Σύστημα Ασφάλισης των Καταθέσεων κλπ. Ε, πρέπει να το κάνουμε. Βέβαια, βλέπουμε διστάμενες απόψεις ανάμεσα στα κράτη Πιστεύουμε όμως ότι πρέπει να προχωρήσουμε μέχρι το τέλος, όπου να έχουμε απόλυτα αμοιβεοποιημένους κινδύνους σε όλη την Ευρωζώνη. Και τμήμα αυτού φυσικά θα είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης των Καταθέσεων. Τα μέτρα αυτά θα ε, διασφαλίσουν ε, την ακεραιότητα της Ευρωζώνης ε, τα επόμενα χρόνια. Αν ε, όμως ε, περάσουμε σε έναν ε, φαύλο κύκλο, αυτό θα, δεν θα είναι καλό και θα πρέπει να συνομιλήσουμε με ως τον τομέα αυτών. Ακόμα και αν έχουμε ένα καλάθι συναλλαγμάτων, αν υπάρχει ένα ασθενές συνάλλαγμα, αυτό μπορεί να επηρεάσει όλη την κατάσταση και θα επιλέξει κανείς να επενδύσει σε μια πιο ασφαλή ζώνη. Ανησυχώ λοιπόν ότι θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις αν δεν ε, προσέξουμε ιδιαίτερα το θέμα αυτό και εάν δεν προσπαθήσουμε απλά να βολέψουμε όλες τις πολιτικές απόψεις, αλλά να ε, φροντίσουμε να έχουμε ακαιρεότητα μιας απόφασης ε, για το μέλλον της Ευρωζώνης. Όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και το κατά πόσο οι τράπεζες είναι κερδοφόρες, ήμουν βουλευτής στην Ιρλανδία επί πολλά χρόνια κατά ένα πολύ δύσκολο χρονικό διάστημα, διότι χρεοκοπούσαν τράπεζες και είχαμε και όλα τα προβλήματα που προκύπτουν από κάτι τέτοιο. Είναι λοιπόν απαραίτητο να είναι κερδοφόρες οι τράπεζες και το γεγονός ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν κλειστεί εντός των συνόρων τους σημαίνει ότι δεν έχουμε πολλές διασυνοριακές τραπεζικές πράξεις. Εάν όμως θέλουμε στα σοβαρά μια ενιαία αγορά θα πρέπει να εξετάσουμε πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε οι διασυνοριακές ασφα... Ε, υπηρεσίες να ε, ε, να συνεχίσουν να διεξάγονται, να έχουμε ένα σύστημα που να μην εμποδίζει τις διασυνοριακές τραπεζικές συναλλαγές. είναι ακόμα και δύσκολο να ε, λάβει κανείς ε, δάνειο από άλλη χώρα. Τέλος, όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, και πάλι, πρόκειται για τομέα όπου κάποιες χώρες έχουν προοδεύσει πάρα πολύ, ενώ άλλες όχι. Άσχετα όμως από το τι πίεση ασκείται στις χώρες για να αντιμετωπίσουν το θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, το θέμα είναι ότι από κοινωνικής πλευράς θα πρέπει να φροντίσουμε αυτούς ε, που χρωστούν όταν τα χρέη αυτά πολλούνται ε, σε επιθετικά ταμεία, σε επιθετικούς οργανισμούς ανάκτησης ε, των χρεών. Και στην Ιρλανδία το είδαμε αυτό. Θα πρέπει να υπάρχει προστασία. Δεν μιλάμε απλά για σολογισμούς, μιλάμε για τις ζωές ε, και τις επιχειρήσεις ανθρώπων. Κάποιες χώρες ακόμη δεν ε, έχουν αντιμετωπίσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, δεν θα επιτρέπεται όμως να πωλήσουν τα δάνεια αυτά ε, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να πωλήσουν τα δάνεια αυτά χωρίς να υπάρξει απαραίτητη προστασία για τους δανειολήπτες. Τα σημαντικά πολιτικά ζητήματα θα στρέφονται γύρω από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης των Καταθέσεων και τα Safe Assets. Ευχαριστώ κύριε Σούρτασον από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Για τον εισηγητή, τους κοιόδρους εισηγητές, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τον κύριο Μάρκες για το σχέδιο εκθεσής του που αναφέρει πολλές σημαντικές πτυχές και όλη η προετοιμασία στις διάφορες συναντήσεις που οργάνωσε ο εισηγητής βοήθησαν πάρα πολύ και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Έχει προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά αυτή η έκθεση. Τώρα, ε, κυρίως μας ικανοποιεί η διατύπωση που μιλάει για κονδύλια προς βιώσιμες ε, ε, επενδύσεις βιώσιμης ανάπτυξης είναι πράγματα τα οποία λαμβάνονται υπόψη και στο θέμα των πλουσιακών στοιχείων και τη σημασία που έχει η προστασία ε, των ε, δανειστών, όπως ε, τα είπε και ο συνάδελφος από το Ρηνιού, για τις ανησυχίες όσον αφορά τις δραστηριότητες του σκιώδου τραπεζικού συστήματος, για την ενίσχυση της ασφάλειας όσον αφορά τραπεζική εποπτεία και για την καταπολέμηση τη συνομοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επίσης, ε, ευχαριστούμε για αυτά που λέει η έκθεση για την ενίσχυση του πυλώνα που αφορά το σύστημα ασφάλιση καταθέσεων. Όμως θα θέλαμε πιο συγκεκριμένε προτάσεις και γι' αυτό και θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες για ε, πρόσφατες περιπτώσεις τραπεζών που φαίνεται ότι από τα στοιχεία που δίνουν οι τράπεζες η αρχή για την εξυγίανση είναι κάτι που παραμένει περισσότερο στα χαρτιά παρά στην πράξη. Έπειτα για τα βιώσιμα δημοσιονομικά θα έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις για δοκιμές όσον αφορά ε, τον άνθρακα και επίσης όσον αφορά την λεγόμενη brown taxonomy, δηλαδή την ταξινόμηση επενδύσεων σε μη, καθαρές, ε, μη καθαρής τεχνολογίας. Θεωρούμε λοιπόν συνολικά ότι το σχέδιο έκθεσης αποτελεί μια πάρα πολύ καλή βάση για να δουλέψουμε απάνω και να περιμένετε ότι θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες για να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Προσβλέπουμε και εμείς σε καρποφόρες συζητήσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Σέντεβαν τώρα, Γκουε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεσή του Ευχαριστούμε και για τι συνομιλίε που είχαμε ω και εισηγητές. Σας ευχαριστώ εκ μέρου τη ομάδα μου. Εδώ λοιπόν σε κάποια πράγματα συμφωνούμε, ιδίω όπω αντιλαμβανόμαστε το θέμα του σκιώδου τραπεζικού τομέα ή το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματο ή τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Είναι σημεία στα οποία μπορούμε να ακολουθήσουμε τη γραμμή του εισηγητή. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά αλλά δεν μπορώ να συμφωνήσω πλήρω με τον ενθουσιασμό σας ε, σε σχέση με τα όσα έχουν επιτευχθεί τα τελευταία δέκα χρόνια για να ε, δούμε πώς ξέσπασε η χρηματοοικονομική κρίση και πόσο σταθερότερος είναι τώρα ο τομέας αυτό σε σχέση με το τι συνέβαινε πριν από μια δεκαετία. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία δεν αντιμετωπίστηκαν πολιτικώς και είναι δική μα δουλειά να αναλάβουμε δράση. Ιδίω με συγκεκριμένε προτάσεις στην περίπτωση των too big to fail ή του διαχωρισμού εμπορικών επενδυτικών δραστηριοτήτων στις τράπεζες ή το τι γίνεται με τους Ευρωπαίους πρωταθλητές, τις τεράστιες αυτές τις ε, τράπεζες που έχουν συσσωρεύσει δραστηριότητες. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορεί η συγκέντρωση κεφαλαίων να μην, δημιουργήσει, ε, να μην δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα. Υπάρχει πολύ πολιτική συζήτηση γι' αυτό. Τι περιουσιακά στοιχεία μπορούν να διαθέτουν οι τράπεζες, πόσα και όσα έχουμε αποφασίσει ως τώρα, εμένα δεν μου φαίνεται ότι αρκούν. Εφόσον προκύψει μια νέα οικονομική κρίση, αυτό και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το νέο σύστημα εξυγίανσης θα δημιουργήσει προβλήματα. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε την εξέλιξη και να μπορούμε να παρέμβουμε στο μέλλον. Ε, η ε, Φόρες στο μέλλον θα πρέπει να ε, μην επιτρέψουν ε, να έχουμε τέτοια προβλήματα με τον τραπεζικό κλάδο όπως είχε συμβεί στο παρελθόν. Και θα πρέπει να υπάρξουν τέτοιε διευθετήσει, ώστε μικρέ τράπεζε, αυτέ που έχουν τι αποταμιεύσει των πολιτών, να μπορούν να προστατευτούν. Να μην πρέπει να πληρώσουν το τίμημα. Θα πρέπει λοιπόν κάπω τα πράγματα να τα εξορροπήσουμε σωστά. Και γι' αυτό θα κοιτάξουμε ω και ο να συνεισφέρουμε επικοδομητικά στην όλη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. So we have, uh, Καλώς. Για Eye, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Ρένα Μάρκες, παρακαλώ, η πρώτη ερώτηση στο Eye. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να ξεκινήσω χαιρετώ, χαιρετίζοντας τις προσπάθειες του εισηγητή για την έκθεσή του τον ευχαριστούμε, τον ευχαριστούμε για την ε, διξοδικότητα της όλης έκθεσης και για τις ε, πολύ κέρυες παρατηρήσεις του, τις οποίες αυτή τη στιγμή συζητούμε. Η έκθεση αυτή είναι πολύ θετική και προς τη σωστή κατεύθυνση. Ήθελα να θυμίσω, όπως ήδη υπόθηκε, ότι πρέπει να αναζητήσουμε να εντοπίσουμε μάλλον τη σημασία τη ε, συμπεριφορά τη Οικονομική και Νομισματική Ένωση, ιδίω σε μια χρονική συγκυρία, όπου όταν εγκρίθηκε η δήλωση τη Ρώμη ε, ω συμπλήρωμα τη συνθήκη τη Ρώμη πριν από δύο χρόνια, ο Πορτογάλος Πρωθυπουργό είπε ότι θα προσυπέγραφε αυτή τη δήλωση αν υπήρχε κείμενο της δήλωσης με ρητές αναφορές την συγκεκριμένη συμπεριφορά που αναμένουμε από την Οικονομισματική και Νομισματική Ένωση. Εδώ λοιπόν ήθελα πολύ συγκεκριμένα να αναφερθώ σε μια γενική παρατήρηση σε σχέση με τη σταθεροποίηση. Ένα μηχανισμό σταθεροποίησης. Θεωρώ ότι εδώ πρέπει να είμαστε πιο απαιτητικοί και μπορούμε να είμαστε πιο απαιτητικοί ήδη από αυτή την έκθεση, δίνοντας ε, έμφαση στην ε, ιδιότητα τη σταθεροποίησης που αναφέρεται εδώ, λαμβάνεται υπόψη, αλλά να είμαστε κάπως πιο συγκεκριμένοι στην αντασφάλιση για την απασχόληση από τη μία και από την άλλη την ανάγκη να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την εξέβρεση εργαλείων ε, σύγκλησης, το BIC ας πούμε όπου έχουν γίνει κάποια βήματα πρόοδου στο επίπεδο του Συμβουλίου. Αλλά πάνω απ' όλα σημαντικό είναι να προχωρήσουμε με το μηχανισμό της σταθεροποίησης υπό την έννοια Τη αντιμετώπιση αντίξων συνθήκων που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη, ώστε να μην τίθεται να αμφιβόλο η επενδυτική τους ικανότητα. Αυτό για μένα είναι το σημείο κλειδί που θα πρέπει να ε, αποσαφηνίσουμε εδώ σε σχέση με τη λειτουργία της σταθεροποίηση. Ευχαριστώ πολύ. Very ε, ε, ευχαριστώ πολύ, κύριο Σίλβα Περέιρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον ε, συνάδελφο Μάρκε για την εξαιρετική έκθεση που υπέβαλε σε σχέση με την ολοκλήρωση τη Τραπεζική Ένωση. Ε, με πολύ καλή ανάλυση και εντοπισμό των προβλημάτων ε, διότι είναι πολύ καλή η αντίληψή του για τις προκλήσεις που θα έχει να αντιμετωπίσει η Τραπεζική Ένωση στο μέλλον γνωρίζουμε την ατζέντα, το πρόγραμμα για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης έχει οριστεί με ιδιαίτερη λεπτομέρεια, κατά λεπτός θα έλεγα. Οπότε η έκθεση ε, κοιτάζει τις θετικές πολιτικές δηλώσεις ως προς την επίτευξη της τραπεζικής ολοκλήρωσης. Ιδίως ως προς το ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης των καταθέσεων και τη λειτουργία του ενιαίου μηχανισμού ε, εξηγένση καθώς και του μηχανισμού σταθερότητας. Εφόσον ε, εντοπίσουμε αυτούς τους πυλώνες που λείπουν από την Τραπεζική Ένωση θα μπορούμε να προχωρήσουμε. Να θυμηθώ εδώ μια ταινία που αναφέρεται η γέφυρα που έλειπε στα ελληνικά γέφυρες του Μάρντισον. Εδώ λοιπόν Έχουμε κάνει μια συζήτηση πολύ ε, εντατική για τη διαφορά συστημικών κινδύνων και μείωσης κινδύνων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι ποτέ δεν ε, έχει να αντιμετωπιστεί αρκετά κίνδυνοι, οπότε δεν μπορούν και να κατανεμηθούν διαφορετικά. Ε, με την επιφύλαξη λοιπόν εδώ των οικονομικών ευθυνών που θα πρέπει να αναλυφθούν εδώ, να θυμηθώ ότι στην προηγούμενη θητεία εγκρίναμε εδώ σε αυτό το Ευρωκοινοβούλιο ένα νομοθετικό πακέτο πολύ απαιτητικό για το χρηματοοικονομικό σύστημα. Με την ε, άποψη ότι αυτό το βήμα έλειπε για να προχωρήσουμε στην Τραπεζική Ένωση. Εδώ λοιπόν ήθελα να ρωτήσω στο, τον εισηγητή βάσει της αξιολόγησης που έκανε πώς μπορούμε να βρούμε κατάλληλες προϋποθέσεις, ε, αρκετές προϋποθέσεις, για να φτάσουμε στην ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και τι πρέπει να κάνουμε για ένα νέο πακέτο μείωσης του κινδύνου, εφόσον κρυφεί απαραίτητο. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα λόγο στον εισηγητή για τρία λεπτά για την απάντησή του. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια, για τις ερωτήσεις. Πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέρουσες όλες οι προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι από αυτά που άκουσα, νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε στη βάση για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, όπως επίσης και για κάποιους κινδύνους που προέκυψαν όλα αυτά τα χρόνια. Και όπως ακούσαμε μόλις τώρα, είχαμε μείωδο, μείωση κινδύνων και επιμερισμό των κινδύνων χάρη σε αυτή τη διαδικασία. Συνεπώς, Κάποια από τα θέματα που θίξατε εξαιτία των κανόνων που ισχύουν για τις εκθέσεις αυτές, ε, τα είπαμε στις ε, συνεδριάσεις μας, προσπάθησα να τα συμπεριλάβω, αλλά θα έπρεπε να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο και να διατυπωθούν ακόμα καλύτερα στην τελική έκθεση. Είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσουμε επ' αυτού. Τώρα, η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης δεν πρόκειται μόνο για το ΕΝΤΙΣ την ασφάλιση καταθέσεων ή τη σχέση δημοσίου χρέους με τράπεζες. Πρόκειται επίσης και για την συγκέντρωση οφειλών στα χαρτοφυλάκια τραπεζών. Πάντως, επί του παρόντος, τα βήματά μας πρέπει να είναι πολύ καλά ισορροπημένα και συμφωνώ ότι τα επόμενα βήματα θα πρέπει να έχουν και τον επιμερισμό των κινδύνων ως ε, στοιχείο. Είναι πράγματα που εγκρίθηκαν και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που ήταν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση υπέρ του ΕΝΤΙΣ, της ασφάλισης καταθέσεων, έτσι κι αλλιώς και ίσως κάνουμε κάτι παραπάνω. Δηλαδή τα καθεστώτα ρευστότητα ίσως και αυτά κάπως να τα ενοποιήσουμε περισσότερο. Και υπάρχει και κάτι άλλο που είναι σημαντικό. Η εμπιστοσύνη. Χρειάζεται ε, περισσότερη εμπιστοσύνη στις αρχές, ώστε αυτή η τραπεζική ένωση να μας απαλλάξει από τα μέχρι τώρα προβλήματα. Σίγουρα πολλούς δρόμους μένει να καλύψουμε, αλλά υπάρχει ελπίδα. Από τις τελευταίες ευρωεκλογέ έχω την αίσθηση ότι πήραμε ένα σαφές μήνυμα ότι πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο. Δεν μπορούμε να εμποδίζουμε, να κρύβουμε τα πιο σημαντικά ζητήματα. Θέλουμε την Οικονομική και Νομισματική Ένωση και την ολοκλήρωσή της, αλλά η Τραπεζική Ένωση είναι κάτι βασικό που μπορεί να μας βοηθήσει στην εκπλήρωση των ονείρων μας. Ωραία, περιμένω τις τροπολογίες και πιστεύω πραγματικά ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία για την τελική έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Υπενθυμίζω ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την έκθεση αυτή. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 13 Δεκεμβρίου. Θα εξετάσουμε τις τροπολογίες 22-23 Ιανουαρίου και θα ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή μας ή στις 17 ε, ή στις 18 Φεβρουαρίου. Οπότε το Μάρτιο μπορούμε να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια, το Μάρτιο του 2020. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Ωραία, οπότε νομίζω ότι τώρα ε, μπορούμε να κηρύξουμε την λήξη της συνεδρίασής μας και να συνεχίσουμε με τη συνεδρίαση των συντονιστών. Οπότε οι υπόλοιποι που βρίσκονται στην αίθουσα και που δεν πρέπει να είναι εδώ στη συνεδρίαση των συντονιστών να αποχωρήσουν. Ευχαριστώ.